Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε δύο σημαντικές ακροάσεις σήμερα. Ξεκινάμε την ημέρα σε διάταξη, δεν ξέρω αν έχετε σχόλια, αλλιώς μπορούμε να την εγκρίνουμε. Έχετε σε 19 γλώσσες ε, διερμηνία και αύριο σε 16. και βέβαια μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της 24ης ε, Μαΐου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ελήψει σχολείων θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τα σχόλια μα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Κρίστοφ Γκάους, ο οποίος είναι επικεφαλής του το ελέγχου εκπομπών και δοκιμασίας αυτοκινήτων από το ΑΝΤΑΚ, το γερμανικό, τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου. Χαιρόμαστε που είστε εδώ παρόν. Φυσικά εκπροσωπείτε τη μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτου στην Ευρώπη με έδρα στο Μόναχο και συμβουλεύετε τους ε, οδηγούς για όλα τα θέματα αυτοκίνησης και επίσης έχετε και το εργαστήριο για τον έλεγχο και τις δοκιμασίες αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά τα καυσαεριά τους. Όπως πάντα αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα και 40 λεπτά σε δύο γύρους, αλλά θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Γκάους, ο οποίος έχει το λόγο για 10 λεπτά κατά μέγιστο. Σας ευχαριστώ κυρία Φανμπρέντ. Κρίστοφ Γκάους λέγομαι. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω γερμανικά, γιατί έτσι μπορώ να δώσω και πιο λεπτομεριακές απαντήσεις στα ερωτήματα. Να σας παρουσιάσω καταρχήν το ADAC, τη λέξη αυτοκινήτων. Ξέρετε ότι είναι, είναι ο δεύτερος, η δεύτερη μεγαλύτερη λέξη στον κόσμο. Έχουμε 19 εκατομμύρια μέλη στη Γερμανία και ο στόχος της εργασίας μας είναι μεταξύ άλλων να δώσουμε στον την καλύτερη πληροφόρηση στα μέλη μας για τεχνικά θέματα και επίσης να τους συμβουλεύσουμε και για αγορές αυτοκινήτων. Γι' αυτό ε, δοκιμάζουμε περίπου 150 οχήματα κάθε χρόνο και μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες περιλαμβάνονται και οι δοκιμασίες για τις εκπομπές αλλά φυσικά και πολλά άλλα στοιχεία. Έχουμε το κέντρο μας ε, έξω από το Μόναχο, βλέπετε εδώ πέρα στο, στην εικόνα το τεχνικό κέντρο του ADAC. Ε, Έχουμε περίπου 200 εργαζομένους στο κέντρο δοκιμών μας και κάνουμε δοκιμές σύγκρουσης, δοκιμές ε, οδήγησης στο δρόμο, κάνουμε και άλλες βέβαια τεχνικές ε, δοκιμασίες όπως ε, παραδείγματος χάρη για τα αυτοκίνητα ε, περιπολίας στους δρόμους εκεί γίνεται η εκπαίδευση των οδηγών τους και εκεί προσαρμόζονται τα αυτοκίνητα τα οποία είναι υπεύθυνα για περιπολίες στους δρόμους και φυσικά έχουμε αυτή τη συνεργασία και με, φορούς, με φορείς που ενδιαφέρονται για αυτές τις δοκιμασίες. Έχουμε 160 ε, εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται με, τα, με τις δοκιμασίες αυτές. Κάνουμε δοκιμές επί τη βάση και συμφωνιών με διεθνείς εταίρους. Βλέπετε τώρα τα λογότυπά μας που είναι κάπως δύσκολα να τα διαβάσετε αλλά βλέπουμε, βλέπετε εκεί ότι υπάρχουν εκπρόσωποι από διάφορες ε, οργανώσεις όπως είναι το ATRC που είναι η Διεθνής Ένωση Δοκιμασίας για τους Καταναλωτές. <clears throat> Όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία μας και έχουμε και συνεργασία σε θέματα έρευνας με τις διάφορες εθνικές και τοπικές αρχές, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και με την Ομοσπονδιακή ομοσπονδιακές αρχές της ε, Γερμανίας. Γιατί λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλος δώρος γύρω από τον κινητήρα diesel. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία φυσικά σας ε, είναι απόλυτα γνωστά, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα στοιχεία. Καταρχήν έχουμε ε, εργαστηριακές δοκιμές οι οποίες γίνονται στην Καλιφόρνια, στο California Air Resources Board, στο CARB και εκεί έγιναν οι πρώτες δοκιμές οι οποίες κατέληξαν, βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια τώρα, έχετε τον Αμερικάνικο κύκλο, ο οποίος είναι γνωστός ως FTP75. Και οι οριακέ τιμέ για, αυτόν τον, για αυτή τη δοκιμασία είναι η πράσινη γραμμή. Αλλά βλέπετε ότι με τους ευρωπαϊκούς κύκλους ε, δοκιμής είναι πολύ χειρότερες οι αποδόσεις τους επί τη βάση του ευρωπαϊκού κύκλου, ενώ οι αμερικάνικες δοκιμές είναι αυστηρότερες. Και ακόμα και αν έχουν προσαρμοστεί αυτά τα οχήματα στους αμερικανικούς τρόπους δοκιμασίας, είναι παράξενο αυτό το αποτέλεσμα. Έχετε στη συνέχεια το το, τις δοκιμές που έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βυργινίας που έκανε δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες, όχι με τα ίδια αυτοκίνητα, αλλά σε συγκρίσιμες συνθήκες. Προσπάθησαν να δουν τι γίνεται όταν κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο σε πραγματικές συνθήκες με τις εκπομπές. Κάνανε ένα κύκλο, ένα σιρκουί ε, στο Σαν Φρανσίσκο. Και εδώ βλέπουμε πάλι στις, ε, στην επόμενη διαφάνεια Έχουμε τα τρία αυτοκίνητα A, B και C και βλέπουμε τις ε, τιμές αυτές που κανονικά θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από την πράσινη γραμμή που είναι το όριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπετε μετά τις πραγματικές εκπομπές οι οποίες είναι φυσικά πολύ υψηλότερε. Και βλέπουμε λοιπόν που βρίσκεται το πρόβλημα ήδη για μας το αντεατσέ, όλα αυτά δεν μας φαίνονται ότι είναι μια τεράστια ε, έκπληξη. Εμείς έχουμε τα δικά μας εργαστήρια από το 1979 και κάτω από διαφορετικές συνδίκες μπορούμε να κάνουμε και δοκιμές εκτός ε, κύκλου, που δεν είναι η κύκλη η επίσημη για τις δοκιμές, αλλά ο στόχος μας είναι στις δοκιμές αυτές που κάνουμε το αντεατσέ, να δώσουμε στα μέλη μας πληροφόρηση για τις πραγματικές τιμές εκπομπών των αυτοκινήτων. Επομένως θέλουμε απλώς να δώσουμε συμβουλές στα μέλη μας για την κατανάλωση των οχημάτων, γιατί αυτό είναι το πρώτο θέμα που τους ενδιαφέρει. Πόση βενζίνη, πόσο δίζελ καταναλώνει το αυτοκίνητο που έχουν αγοράσει, αλλά φυσικά έχουμε μετρήσει και τις εκπομπές των ε, ρήπων και έχουμε κάνει αυτές τις λεγόμενες οικολογικές δοκιμές όπου ε, καταμετρούμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και του αζότου και συνολικών υδρογονοανθράκων. Κάνουμε λοιπόν αυτές τις ε, δοκιμές, δεν παρουσιάζουμε βέβαια τις ε, λεπτομέρειες των ε, δοκιμών μας, αλλά δίνουμε μια γενική αξιολόγηση για κάθε όχημα. Και εδώ κάναμε μια δοκιμασία, κάναμε μια αξιολόγηση το τεστ μας έχει να κάνει με τρεις κύκλους οδήγησης. Κάνουμε καταρχήν κάτι το οποίο είναι σχεδόν ο επίσημος ε, κύκλος για την έγκριση. Ακολουθούμε τις ε, ενδείξεις που υπάρχουν για την αλλαγή ταχυτήτων από τον κατασκευαστή, αλλά κάνουμε και δύο δοκιμασίες εκτός κύκλου, ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε το 2012 για τους συνολικούς ε, ε, υδρογονάνθρακες και βλέπετε την ε, κόκκινη γραμμή ενώ η μπλε γραμμή είναι η επίσημη. Έχουμε λοιπόν ένα, την εφαρμογή ενός νέου κύκλου με ένα παγκόσμιο πρότυπο και χρησιμοποιούμε εδώ την εκκίνηση με τον κινητήρα εν θερμό, όχι εν, εν Και έχουμε λοιπόν ε, τις πληροφορίες για, το, για να έχουμε πληροφορίες τι γίνεται στο δρόμο. Έχουμε ένα κύκλο σε που περιλαμβάνει και αυτοκινητόδρομο. Ε, και μπορούμε να δοκιμάσουμε τι γίνεται με τους διάφορους τρόπους καταμέτρησης. Και όχι μόνο το VL ΤΕΣΕ και τον ΕΦΤΣ. Και έχουμε λοιπόν επίσης αναπτύξει μαζί με την ΤΥΦ την υπηρεσία ελέγχου των αυτοκινήτων ε, στην ε, Βάδη Βιρτεβέργη και στην Βόρεια Γερμανία. Έχουμε αναπτύξει κοινέ δοκιμές αυτοκινήτων με τρία αυτοκίνητα τα οποία έχουμε δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες. Είναι ε, αυτοκίνητα diesel τα οποία συμμορφώνται με το πρότυπο Euro 6 και βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα. και έχουμε καταλήξει εδώ σε μια ε, συνολική αξιολόγηση για 40 αυτοκίνητα diesel και βλέπουμε τον παράγοντα απόκλησης ή τον παράγοντα συμμόρφωσης όπως αναφέρεται σε πολλές περιπτώσεις ο οποίος ε, υποτίθεται πρέπει να είναι στα 2,1. Ε, Αν δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα οχήματα αυτά, υπάρχει ο παράγων αυτός απόκλησης από το VLTC, από τον Παγκόσμιο Κύκλο Δοκιμασίες. Βλέπετε λοιπόν τα οχήματα αυτά, τα οποία έχουν ένα υψηλότερο παράγοντα συμμόρφωσης. Και εδώ όμως μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και με τα δικά μας ε, ε, τεστ υπάρχουν πολλά οχήματα τα οποία ξεπερνούν τα όρια αυτά. Κάποια έχουν ε, περάσει με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο τον, ε, το τεστ αυτό. Εδώ σας παρουσιάσουμε τρία οχήματα, τη Mazda 6, την BMW 320 και το Passat Setzet και βλέπετε ότι σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης υπάρχει Φυσικά περιμένει κανείς ε, να είναι πιο ψηλές οι τιμές και υπάρχει μια σημαντική απόκληση, οπότε πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο φάσμα αποκλήσεων που ίσχυε και για οχήματα της κατηγορίας Euro 6 και επίσης και η κατηγορία Euro 5 ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και εμείς έχουμε δημοσίευσει όλα αυτά τα στοιχεία. Και εδώ βλέπετε πάλι μια κατάταξη οχημάτων επί τη βάση των ε, παραγόντων εκπομπών. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο σε σχέση με τους ε, παράγοντες αυτούς. Η... Τα κίτρινα σημεία είναι αυτά που αφορούν τα ευρώ 5 και ευρώ 6. Από τη μία πλευρά, μάλλον στον ε, στον άξονα των Χ βλέπετε την ταχύτητα και στον ε, άξονα των Ψ βλέπετε τις εκπομπές ε, οξύδια του αζότου. Και αυτό το οποίο μπορεί να, να δει ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές και σε χαμηλές ταχύτητες και σε υψηλές ταχύτητες όπου οι εκπομπές είναι πολύ πιο ψηλές από τις οριακές τιμές οι οποίες θα έπρεπε να ισχύουν για το, τα ευρώ 6 και, ε, και 5. Αυτό το είδατε για το Passat, αλλά παρόμοια είναι η κατάσταση και με την Mazda και με την BMW. Ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το κάθε όχημα, σε όλες τις περιπτώσεις είναι φανερό ότι χρήζουν βελτιώσεως, αν είναι να περιληφθούν από την, να περιληφθούν στα πρότυπα Euro 5 και Euro 6. Και εδώ βλέπετε διάφορες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών. Έχω ήδη αναφέρει αυτό σε προηγούμενες ακροάσεις και δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς περιμένω να θέσετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα ξεκινήσουμε με τους δύο εισηγητές. Ο κύριος Σάλμπα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε λοιπόν. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις τις οποίες μας δώσατε εδώ σήμερα. Το πρώτο είναι η... Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε εγώ δεν είμαι τεχνικός και θα ήθελα να το εξηγήσουμε. Οι δοκιμές τις οποίες κάνετε εσείς είναι αποκλειστικά εργαστηριακές ή γίνονται επίσης ε, και δοκιμές ε, με κινητά συστήματα ελέγχου. Dies sind bis jetzt nur Labortests. Εμείς αυτά τα οποία παρουσιάζω εδώ είναι μονάχα τεστ στο εργαστήριο. Εμείς έχουμε δει βέβαια ότι εκτός του επισήμου κύκλου, όταν μετρήσουμε εκτός του επισήμου κύκλου, αυξάνονται οι εκπομπές. Αλλά πριν από δύο χρόνια σκεφτήκαμε να έχουμε ένα σύστημα κινητό, ένα σύστημα PEMS, το οποίο να ε, ακολουθεί το αυτοκίνητο στον δρόμο και υπάρχουν πολλές οργανώσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να αγοράσουν τέτοιες συσκευές και έχουμε μια τέτοια ε, συσκευή και γι' αυτό είναι η πρόθεσή μας να κάνουμε και περαιτέρω δοκιμασίες με κινητά συστήματα μέτρησης ε, ρήπων. Ευχαριστώ κύριε Κάουσο. Είπατε ότι εδώ και δύο χρόνια περίπου ξεκίνησατε να χρησιμοποιείτε αυτά τα κινητά συστήματα. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι τρέφατε κάποιες υποψίες, ότι κάποιοι κατασκευαστές είχαν σαν σχέδιο να έχουν τακτικές για, την, ε, ε, για να ακυρώνουν την, ουσιαστικά τη μέτρηση που γίνεται επισήμω ή το κάνατε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια υποψία. Δεν είχαμε κάποια υποψία ότι είχαν γίνει χειραγωγήσεις. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το διακριβώσουμε με τις δικές μας δοκιμασίες αν υπάρχει κάποια χειραγώγηση. Όχι, απλώς βλέπουμε ότι είναι διαφορετικές οι πραγματικές εκπομπές από αυτές που μετράει κανείς στο εργοστήριο. Αυτό μπορεί να είναι και αντικειμένο, είναι απαραίτητο μάλλον ένα αποτέλεσμα χειραγώγησης, αλλά μπορεί να είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σχεδίαση των κύκλων. Δεν είναι κάτι το οποίο αδίδυτα σημαίνει ότι είναι μια χειραγώγηση. Απλώς αυτό το οποίο για μας ήταν σημαντικό ήταν ότι διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούν μάλλον να καταμετρηθούν όλες οι εκπομπές στο εργαστήριο και γι' αυτό πρέπει να τις μετρήσουμε και με άλλους τρόπους. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, θα θεωρήσει υποχρεωτικές τις δοκιμές ε, τα τεστ σε πραγματικές συνθήκες. Ο υποχρεωτικός αυτός χαρακτήρας θα αλλάξει κάπως τον τρόπο που προσμετράτε. Θα αξιολογήσετε, εν πάση περιπτώσει, τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να γίνει υποχρεωτικό το σύστημα και σε ποιο βαθμό θα αλλάξει ο τρόπος που συνεργάζεστε. Zunächst unterstützen wir εμείς υποστηρίζουμε απόλυτα τη νέα οδηγία για να γίνει υποχρεωτική η δοκιμασία στον δρόμο και να μετρούνται εκεί στον δρόμο. Το έχουμε ήδη προτείνει στο παρελθόν, ακόμα και όταν δεν είχαμε εμεί κάποια δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο και δεύτερον πρέπει να παρουσιαστεί η πραγματική κατάσταση για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Και ήδη εμείς προετοιμαζόμαστε για να προχωρήσουμε ώστε στις οικολογικές μας δοκιμές να γίνονται περισσότερες πιο επακριβείς ε, μετρήσεις και επίσης χρειάζεται να υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις τιμές οξυδίου του αζότου και γι' αυτό είναι απαραίτητη και η κύκλη δοκίμης σε πραγματικές συνθήκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκάους. Um, going through your uh, written answers, I... Βλέποντας και τις γραπτές σας απαντήσεις, βλέπω ότι ασκείται κριτική απέναντι στις αυτοκινητοβιομηχανίες, προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Στην ερώτηση υπαρίθμε νέα λέτε και ότι η εισαγωγή των κανόνων εκπομπής 6, ε, Euro 6, δεν ήταν κάτι το οποίο βοήθησε ή οδήγησε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να λειτουργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Είναι μια σκληρή κριτική και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λήψη αποφάσεων συνειδητοποιούσαν τις τεράστιες αποκλήσεις. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Εγώ ξέρω ότι το Άντακ είναι μια λέσχη ιδιαίτερα σημαντική που επηρεάζει πολλά στη Γερμανία και οι Γερμανοί είναι ικανότατοι στο να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Μπορείτε να μας πείτε ε, τι συνέβη όταν συζητήσατε τα ευρήματα των δικών σας δοκιμών με τις γερμανικές αρχές. We sometimes discussed uh, this, uh, uh better speak in German. We are... Ναι, έχουμε στα γερμανικά. Έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα θέματα με τις αρμόδιες αρχές Μα και οι αρχές τα ξέραν αυτά τα θέματα. Και από τα ίδια τα Υπουργεία, από το ίδιο το Υπουργείο, υπήρξε η έκφραση της θέλησης να εξελίξουμε διαφορετικές μεθόδους ε, δοκιμασίες. Γι' αυτό υπήρξε η υποστήριξη και από το Υπουργείο να αναπτύξουμε δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες. Και εμείς φυσικά θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. παρά την στάση αυτή του Γερμανού Υπουργού, του Υπουργείου, χρειάστηκε πάρα πολύ καιρός, χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί. Και δεύτερον, συζητήσατε ποτέ μαζί τους κάποιες διαδικασίες επί παραβάση βάρος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Κάτι δηλαδή παραπέρα από την απλή βελτίωση του συστήματος κάτι το οποίο να διευκολύνει και την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος. Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων <clears throat> έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει με το, με το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα γιατί σε πολιτικό επίπεδο δεν προχωρήσαν τα θέματα αυτά επαρκώς και δεν έγινε αυτό το οποίο εμείς ε, θα επιθυμούσαμε να γίνει το ταχύτερο δυνατό, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Και από την πλευρά των κατασκευαστών βλέπουμε ότι οι κατασκευαστές θέλουν να βελτιώσουν τα οχήματά τους, αλλά αυτό το οποίο κάνουν είναι μονάχα αυτό το οποίο είναι αποτέλεσμα μεγάλης πίεσης. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα για τη μείωση των ρήπων. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι, ότι όταν κάνουμε ένα ε, αυστηρότερο τεστ στην αρχή μας κοιτάνε λιγάκι στραβά, μας λένε ότι αυτό θα είναι πολύ πολύ δάπανο λοιπά, Αλλά σιγά σιγά ε, με το διοξείδιο του άνθρακος όταν ετέθη η έμφαση στη μείωση του μέσου όρου εκπομπή διοξείδιου του άνθρακος από το συνολικό στόλο αυτοκίνητο παραγύρα κατασκευαστή, είδατε ότι ανταποκριθήκανε. Μια οργάνωση σαν τη δική σα, τόσο σημαντική στη Γερμανία, υποθέτω ότι θα έχει καλές σχέσεις και με τους μεμονωμένους υπαλλήλους ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και πολλές ανεπίσημες επαφές. Εσείς σε επίπεδο ανεπίσημο συνειδητοποιήσατε ποτέ ότι κάποια μέτρα στην ουσία δεν ε, επετράπει να ληφθούν από κάποιους υψηλά στην ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης. Έχετε την αίσθηση αυτή. Και σε σχέση τώρα με τις δοκιμές σύγκρουσης, αν είχατε την αίσθηση ότι δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο, θα επιτρέπατε να συνεχιστεί να γίνεται κάτι τέτοιο για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη τουλάχιστον με το θέμα των εκπομπών, των δοκιμών για τις εκπομπές. Το δικό μας καθήκον καταρχήν είναι να κάνουμε δοκιμές για να συμβουλεύουμε τα μέλη μας. Είμαστε σύμβουλοι των μελών του ΑΝΤΑΤΣ και φυσικά προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των ε, ε, μελών μας, αλλά δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να τα κάνουμε όλα. Γι' αυτό εστιάζουμε περισσότερο στην παροχή συμβουλών. Χωρίς να υπάρξουν πολιτικές ε, αποφάσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και δεν ξέρω γιατί δεν έχουν ληφθεί οι αντίστοιχε ε, αποφάσεις. Εμείς πάντα έχουμε όμως επαφές με τους αξιωματούχους του αρμόδιου Υπουργείου στη χώρα μας. Γκυζίκης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γκάους πάρα πολύ. Μιλήσαμε για τους νέους κύκλους, το VTLC και το NEDC. Εσείς μιλήσατε για το οικολογικό, οικολογική δοκιμασία που είναι σημαντική για τους καταναλωτές. Μερικές φορές φοβάμαι ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται. Κανείς δεν ξέρει. Μήπως θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κοινά πρότυπα για να μπορούμε να συμφωνούμε για τη βάση υπολογισμού. Και μετά από αυτό θέλω να πω το εξής, ως εκπρόσωπος του ΑΝΤΑΤΣ, πώς βλέπετε εσείς το μέλλον του κινητήρα Diesel. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πάντα ανταγωνιστικός αυτός ο κινητήρας Diesel. Ξέρουμε ότι έχουν ληφθεί ήδη κάποια μέτρα. Εάν πραγματοποιηθούν όλα αυτά, μπορεί να είναι καθαρός ο κινητήρας και επομένως ανταγωνιστικός μπορεί να έχει πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο και έτσι μπορεί να βοηθήσει και την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Προφανώ θα γίνει πιο ακριβώ ο κινητήρα με τη μείωση των εκπομπών, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό σε επίπεδο τεχνικό και επομένω <clears throat> τουλάχιστον στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, ίσω όχι στα μικρότερα αυτοκίνητα, έχει πάντα δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικό αυτό ο κινητήρα, ο δίζελ. αλλά θα οδηγήσει αυτό σε πρόβλημα αν τα μικρά αυτοκίνητα γίνουν πολύ πιο ακριβά και δεν θα είναι προσιτά στους ε, καταναλωτές. Θα υπάρχει δυνατότητα τότε τα μικρά αυτοκίνητα να έχουν την κατάλληλη τεχνολογία για την μείωση των εκπομπών. Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του αυτοκίνητου, περισσότερο με το μέγεθος του κινητήρα, με, από τα από το 1,6 από, το, από τα 2 λίτρα το κινητήρα δίζελ πάντα έχει τη δυνατότητα να, επιβιώσει. Αλλά για τους κινητήρες που είναι 1-1,2 παραγωγικά λίτρο, νομίζω ότι η τεχνολογία των κινητήρων βενζίνης είναι πιο προχωρημένη και μάλλον θα πάρει τον κυρίαρχο ρόλο. Μία ακόμα ερώτηση για την απάντησή σας στην ερώτηση 8 είπατε ή αφήσατε να εννοηθεί καλύτερα ότι με την τεχνολογία PEMS μπορούμε να έχουμε μια αξιόπιστη καταμέτρηση των εκπομπών από τους κινητήρες ε, diesel. Και λέτε ότι υπάρχει ένα, σφάλμα ή μάλλον μια, μια αβεβαιότητα 20-30% στις μετρώσεις των PEMS για κινητή μέτρηση. Εμείς έχουμε το σύστημα αυτό, μόλις ε, το έχουμε εδραιώσει μόνο πρόσφατα. Εμείς ξέρουμε ότι μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τον εργαστηριακό έλεγχο, γι' αυτό οι ε, εργαστηριακές δοκιμασίες θα είναι πάντα απαραίτητες. Όταν εμείς <clears throat> μετράμε με το σύστημα PEMS, θα μπορούμε να παίρνουμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκριθούν με αυτά του ελέγχου στα εργαστήρια. Επομένως, με τον τρόπο αυτό, τα συστήματα PEMS θα μας επιτρέπουν να διασταυρώνουμε καλύτερα τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε και έτσι να μειώσουμε την ε, αβεβαιότητα που έχουμε από τι μετρήσεις. Ξέρουμε ότι ήδη από το περιβάλλον μπορεί να, που γίνεται η, η δοκιμασία μπορεί να υπάρξει αβεβαιότητα. Υπάρχει ένα παράγον διόρθωση για τα οξύδια αζότου, ο οποίο ε, ε, επιτρέπεται σε όλες αυτές τις περιπτώσει. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορούμε με τα συστήματα PEMS να μετρούμε αποτελεσματικά την ε, ισχύ του οχήματος και τη σχέση της ισχύω με, το, με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Νομίζω όμως ότι μπορούμε με τον τρόπο αυτό να κατεβάσουμε τον παράγοντα συμμόρφωση στο επίπεδο του 1,5 με 2. Η κυρία Ρεβό. Ευχαριστώ κύριε Γκάους. Η ΕΝΤΑΚ ανάμεσα στις ευθύνες τις οποίες έχει, έχει επίσης και την προστασία του καταναλωτή. Είναι μία από τις βασικές της αποστολές. Ξέρετε ότι τα νόξ δημιουργούν σε 10.000 πρόωρους θάνατους κατέτος. Αυτό είναι ένα θέμα πάνω στα οποία θα πρέπει να εργαστείτε και σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που ήδη δώσατε τις ε, απαντήσεις 1, 3 και 4 αναφέρεστε σε πολλά θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Καταρχάς επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη να απο δραστηριοποιήσει κανείς το σύστημα ελέγχου των OX, ότι αυτό δεν θα βλάψει δηλαδή τη λειτουργία του κινητήρα και αυτό είναι σημαντικό σαν ενημέρωση. Δεύτερον, η νομοθεσία γενικότερα είναι σωστή και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται σεβαστή γιατί υπάρχουν στις καταγραφές διαφορές στις δοκιμές εργαστήριο και στις πραγματικές ε, δοκιμές, στις δοκιμές πραγματικής χρήσης. Στην ερώτηση 1 λέτε επίσης, στην απάντησή σας, ότι δεν μπορέσατε να βρείτε το λογισμικό το εξαπάτησης που χρησιμοποίησε η ΦΑΟΒΕ και κάθε φορά μας λένε το ίδιο, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοιχνεύσει κανείς τον μηχανισμό ακύρωσης. <clears throat> και για την τέσσερα, την ερώτηση τέσσερα, συμπληρωματική ερώτηση. Πιστεύετε ότι έχει σχέση με το λογισμικό το οποίο ενυπάρχει στους αυτοκίνητα. Πιστεύετε ότι το εμπορικό, εμπιστευτικό, το εμπορικό απόρριτο θα πρέπει να ακυρωθεί έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια που θα επιτρέψει σε όλους τους οργανισμούς να ελέγχουν πραγματικά τον κινητήρα. Γιατί είναι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να γνωρίζουμε αν πράγματι υπάρχει ένας μηχανισμός ακύρωσης του συστήματος ελέγχου καυσαερίων. Αυτός είναι ένας ε, δρόμος που θα μπορούσε να εξερευνηθεί και στην οδηγία υπάρχει η έννοια των βασικών στρατηγικών εκπομπών και των βοηθητικών στρατηγικών εκπομπών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γνωστά, τουλάχιστον στις ε, <clears throat> αρχές για την έγκριση του, η έγκριση τύπου οχημάτων. Δεν μπορεί κανείς να δίδει όλες τις λεπτομέρειες βέβαια, γιατί υπάρχει το απόλυτο αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόημα η πληροφόρηση των υπηρεσιών για την έγκριση τύπου, ώστε να μπορούν να ελέγξουν αυτά τα στοιχεία, ώστε να μπορούν να δείξουν ότι δεν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο μπορεί να παρακάμψει το τεστ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν σε συστηματικό επίπεδο να δοκιμάζουμε και να, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια τέτοια διαφορά. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε λογισμικό υπάρχει θα πρέπει να γίνεται γνωστό στις αρχές για, που είναι για την έγκριση τύπου. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες φαίνεται ότι ένας τέτοιος μηχανισμός για τον έλεγχο των νόξ δεν είναι επαρκής και πρέπει να υπάρξει συνδυασμός δύο συστημάτων. Αυτό ισχύει για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι συχνά στην Ευρώπη. Γιατί? Τι κάνετε σε σχέση με αυτό το θέμα. Εμείς ως Αντάτσε δεν είμαστε αρμόδιοι για να κάνουμε τεχνικές προδιαγραφές. Δεν προτείνουμε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό για τη μείωση των εκπομπών. Εμείς απλώς συμβουλεύουμε τα μέλη μας σε σχέση με όλα αυτά. Στην Ευρώπη υπάρχουν ε, διάφορες τεχνολογίες όπως το EGR και υπάρχει στη συνέχεια ο αποθηκευτής ε, για το, τα οξύδια του αζότου, εδώ τίθεται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κόστος ενός οχήματος. Αλλά προφανώς υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει συνδυασμό των ε, συστημάτων αυτών με την παγίδα για των σωματιδίων κτλ. Και για τα οχήματα βενζίνης θα υπάρξουν και εκεί φίλτρα ε, σωματιδίων. Πιστεύω ότι με μεγαλύτερη πίεση για τα θέματα ελέγχου και μεγαλύτερη αυστηρότητα στου ελέγχου θα βελτιωθεί και η τεχνολογία των οχημάτων και των κινητήρων. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στα δεδομένα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για να έχουμε αξιόπιστες δοπικές και συχνά μπερδευόμαστε στη διαδικασία και δεν καταφέρνουμε να έχουμε σωστά στοιχεία. Όπως και εσείς μας ε, είπατε για την WTKS, την περίπτωση αυτή. Λοιπόν, στη... στους οργανισμούς αυτούς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σωστά οι δοκιμές. Τι εννοείται όμως με τα βασικά στοιχεία. Παραγωγικά για την ε, καμπύλη αλλαγή ταχυτήτων ή κάτι τέτοιο. Σας έδειξα ότι δεν έχω την απαραίτητη τεχνική γνώση νομίζω. Νομίζω ότι κάποια ότι αυτά τα λεγόμενα baseline figures σας δίνουν μια γενική εικόνα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτές οι δοκιμασίες που δεν μπορεί κανείς να παρακολουθείς πώς γίνεται το τεστ, αλλά απλώς βλέπει από έξω τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις δοκιμασίες και συμπληρώνουν τα <clears throat> ερωτηματολόγια. Αυτό το έχουμε αναφέρει και σε σχέση με το παγκόσμιο εναρμονισμένο τεστ για τα ελαφρά οχήματα, το VLTP. Πάντα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ακριβώς το τεστ το οποίο γίνεται. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τα στοιχεία τα οποία δίδονται και να παίρνουμε τους, τα στοιχεία που έχουν γίνει από τους κατασκευαστές σε ένα τεστ με μάρτυρες ή από τις αρχές έγκρισης. Δεν έχουμε λοιπόν την ε, δυνατότητα να δούμε πώς γίνεται και ο έλεγχος παραγωγός χάρη του βάρους ενός οχήματος ή του βάρους ενός παρελκόμενου όταν, ε, όταν δοκιμάζεται αυτό το πράγμα στον έλεγχο. Καλώς. Και για τη διαφάνεια, γιατί και εσείς αναφερθήκατε. Πρόκειται για βελτίωση ώστε να αντιστοιχεί στα πραγματικά αποτελέσματα η δοκιμή στα εργαστήρια. Τώρα, το θέμα της θερμοκρασίας επηρεάζει τις εκπομπές, σωστά. Οπότε θα έπρεπε να επηρεάζεται και η διαδικασία πιστοποίησης. Σύμφωνα με το ρεφ 5 και 6 πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εναρμόνιση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται ή υπάρχουν τεχνικοί λόγοι κατά τη γνώμη σας ώστε κάποια συστήματα να μην μπορούν να περάσουν σε αυτή τη διαδικασία αναρμόνισης. Also in jedem Fall sollten Εν πάση περιπτώσει, οι στρατηγικές για τη μείωση των ε, εκπομπών, το πώς γίνεται δηλαδή η ανακύκλωση των καυσαερίων, αυτό θα πρέπει να γίνεται γνωστό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρουν οι κατασκευαστές εν ώψη της ένδυσης τύπου την τεχνική που χρησιμοποιούν για τη μείωση, είτε πρόκειται για ανακύκλωση καυσίμων ή καυσαρίων ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα το ουσιαστικό είναι να μπορούν να γίνονται τεστ σε πραγματικές συνθήκες με διαφορετικές συνθήκες, ώστε να καλύπτεται ένα φάσμα, ένα ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών και να εξασφαλίσουμε ότι με τη τεχνολογία αυτή, οποιαδήποτε και να είναι, η μείωση των εκπομπών γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και όχι μονάχα σε μία θερμοκρασία ελέγχου. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ για τη διαφάνεια, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Στην έκθεσή σας λέτε ότι απόλυτη διαφάνεια και τα χαρακτηριστικά, την απόδοση καυσίμων και των έλεγχο του καθεστώτος βάσει τον οποίο γίνονται οι δοκιμές πρέπει να εξασφαλίζεται. Υπάρχουν τα τεχνικά δεδομένα βάσει των οποίων θα δίνεται η πιστοποίηση και αν ναι, το VW πόσο έχει αντιμετωπίσει την παρούσα κατάσταση. Εμείς δεν θέτουμε ερωτήματα στο KBI. Παίρνουμε όμως από, το, από την υπηρεσία αυτή για τα ε, αυτοκίνητα οχήματα στοιχεία. Εμείς παίρνουμε και από τους κατασκευαστές στοιχεία για όλα αυτά. Το κατά πόσο τώρα, αν λειτουργεί η ανακύκλωση των, ε, μάλλον η επανακύκλωση των ε, καυσαρίων αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το καταμετρήσουμε. Στον κύκλο NEDC τα πράγματα κανονικά λειτουργούν σωστά, αλλά στους άλλους κύκλους ε, ε, δοκιμασιών βλέπουμε μεγαλύτερες αποκλήσεις. Και υπάρχουν κάποια οχήματα της Volkswagen τα οποία είναι καλά και άλλα είναι λιγότερο καλά σε σχέση με αυτά Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Οι δοκιμές από το 2003 γίνονται σε εσά. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν τα πιο σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τους κινητήρες εκείνη την περίοδο ποια ήτανε. Για τις προδιαγραφές 5 και 6 πιστεύετε ότι βοήθησαν οι δοκιμές να υπάρξει κάποια βελτίωση και αν όχι γιατί. Και αν ναι τι διαφορά έχετε διαπιστώσει στη μέτρηση των εκπομπών βάσει του αρχικού πρωτοκόλλου και του NEDC πρωτοκόλλου. Πιστεύω ότι είναι φανερό ότι επί τη βάση των εκπομπών τα οχήματα ευρώ 4, ευρώ 5, ευρώ 6 συνέχεια βελτιώνεται το προφίλ των εκπομπών. Βλέπουμε και σε επίπεδο ε, σωματιδίων ε, δεν υπάρχει όμως στην πραγματικότητα η μείωση των εκπομπών οξυδίου του, άνθρα, οξυδίου του αζότου στο δρόμο, όπως φαίνεται να υπάρχει στο εργαστήριο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε δοκιμές εκτός κύκλου. Υπάρχουν αυτές, υπήρχαν από την αρχή Αποκλίσεις ανάμεσα στον εργαστηριακό κύκλο και τον πραγματικό κύκλο. Είδαμε διαφορές και με το ΔΕΛΤΣΕ και επίσης υπάρχουν αποκλίσεις αν έχει κανείς τον κλίμα. Ε, έχουμε, έχουμε το, τα τεστ με τον ευρωπαϊκό κύκλο, τον NADC, με θερμό κινητήρα και με τον κλιματισμό να λειτουργεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκπομπή διοξίδιων του αζότου αλλά ακόμα παρουσιάζεται από πολλούς και από τα μέσα ενημέρωσης ότι αυτό είναι πρόβλημα του κύκλου δοκιμών και όχι ένα γενικό πρόβλημα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Heeft πήρατε επαφές, είχατε επαφές με τις γερμανικές αρχές, τη γερμανική οργάνωση, την Deutsche Umwelthilfe για παράδειγμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι δράσεις αναλάβατε εσείς και οι γερμανικές αρχές όσον αφορά τα αποτελέσματα των δοκιμών, γραπτά ενδεχομένως, και ποια ήταν η αντίδραση των γερμανικών αρχών. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες της Ομοσποδιακής ε, Αρχής και των Περιφερειακών Αρχών, σε σχέση μάλιστα και με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε κάποια τέτοια διαφορά. Έχουμε πάντα κάνει κοινέ ε, παρακολουθήσεις ε, σε πραγματικές συνθήκες με την, ε, μαζί με το, την Ομοσπονδιακή Αρχή για τα ε, οχήματα, τα αυτοκίνητα οχήματα. Δεν έχουμε τόσο άμεσες επαφές με την Ένωση, τη Γερμανική Ένωση για το Περιβάλλον και αυτή είναι μια ε, ένωση που εκπροσωπεί διάφορα συμφέροντα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ στα μέλη μας, γι' αυτό παραμένουμε ίσως σε, σε επίπεδο μονάχα συμβουλευτικό αλλά ήδη από τη δεκαετία του 1990 από τις διαφορές, από τις διαφορές που διαπιστώσαμε τότε στις δοκιμές έχουμε ζητήσει πάντα από τους κατασκευαστές να μας δίνουν στοιχεία τα οποία να μπορούν να είναι συγκρίσιμα. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι το να κάνουμε έλεγχο στο δρόμο αυτό είναι μια πολύ καλή ε, τεχνική. Δηλαδή Παίρνουμε αυτοκίνητα, αυτοκίνητα στην, <clears throat> τα οποία είναι ε, μεταχειρισμένα, βλέπουμε κατά πόσο να ανταποκρίνονται στις ε, τιμές οι οποίες ε, είναι οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδου ελέγχους σε πραγματικά αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Σύντομα, παρακαλώ. Ναι, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην βιομηχανία και στα εργαστήριά σας έχει ληφθεί υπόψη. Μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλες διαφορές οφείλονται και σε ε, προβλήματα στα οχήματα. Αν παραδείγματος χάρη ένας καταλήτης δεν λειτουργεί καλά. Και επίσης, αν εμείς είμαστε σε, ένα, σε υψόμετρο, στα 600 μέτρα και δεν ε, αναγνωρίζει το σύστημα ότι είναι διαφορετικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης, εκεί μπορούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Α, εκεί δεν ήταν. Α, εσείς τότε. Καλώ. Κύριε Γκάου. εγώ προσπαθώ να φτιάξω μια χρονική γραμμή για αυτά που λέτε. Είπατε το ECOTES ξεκίνησε το 2003 και είδατε από τότε ήδη ότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, μεγάλες αποκλήσεις. Αλλά ήδη από το 2003 είχατε κάποια, κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχουν διαφορές, ότι μπορούν να υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αλλά φυσικά δεν είχατε τρόπο να ξέρετε αν αυτό είναι το αποτέλεσμα κάποια συραγωγής ή όχι. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Είχαμε αποκλήσει από τότε. Αλλά εμεί δεν κάναμε κάποια οικοτολογία σε σχέση με το αν αυτό οφείλεται στο α ή στο β. Γιατί ακριβώς θεωρούσαμε ότι ήδη υπήρχε αυτή η μεγάλη αδυναμία του κύκλου ε, για τις δοκιμασίες. Εμείς αυτό είχαμε στειάσει περισσότερο την προσοχή μας στην ανάγκη να βρεθούν κύκλοι οι οποίοι θα ήταν πιο ρεαλιστικές. Και αν δεν είναι καλός ο κύκλος, δεν κάνει καλή μέτρηση και των ε, ρήπων. Αλλά η επιστημονική υπηρεσία της Bundestag είχε αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα τα οποία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σε κανονικές συνθήκες. Όταν λοιπόν διαπιστώσατε αυτό το πράγμα, ήταν ήδη το 2003, η επιστημονική υπηρεσία της Bundestag πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2016 έκανε μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε προηγούμενη γνωμοδότηση, εμείς δεν ξέραμε τίποτα και απλώς που ήμασταν στα πλαίσια της, ε, των οικασιών. Ακόμα και τώρα δεν έχει υπάρξει μια ε, σαφήνεια σε σχέση με αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από την επιστημονική υπηρεσία της Bundestag. Επομένως εξακολουθούν να είναι δύσκολα για μας όλα αυτά τα θέματα, αλλά εμείς έχουμε τονίσει ότι υπήρξαν αποκλήσεις. Οπότε Πότε για πρώτη φορά είδατε να υπάρχουν τέτοιες ε, αποκλήσεις σημαντικές και πληροφορήσε το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά εμείς δημοσιεύουμε όλα τα αποτελέσματα των ε, ε, ερευνών μας και ήδη υπήρχε μία σαφής απόκληση για θέματα κατανάλωσης καυσίμων και επίσης και για το διοξείδιο του άνθρακος είχαμε δείξει ότι είναι άλλο το επίπεδο εν εκπομπών από ότι με ψυχρό τον κινητήρα. Αν μπορείτε να μας πείτε πότε ακριβώς έγινε αυτή η συζήτηση με την Ομοσπονδιακή Επιστημονική Υπηρεσία της Bundestag, αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξέρουμε ακριβώς για να έχουμε τη χρονική ε, αλληλουχία των γεγονότων πότε είχατε έρθει σε επαφή με αυτούς και με ποιους. Αν μπορείτε να μου δώσετε τα στοιχεία αυτά γραπτά. Εγώ θα προσπαθήσω. Εμείς ε, έχουμε βέβαια τη βασική μας εργασία που είναι ο έλεγχος των 150 οχημάτων το χρόνο. Όλα τα άλλα ήταν περιφερειακά. Αλλά όταν συναντιέστε με ένα υπουργείο ή με μια επίσημη υπηρεσία, κάπου υπάρχει ένα ίχνος του αν έχει γίνει αυτή η, η συνάντηση. Θα πρέπει να δω πόσο παλιά φτάνουν τα αρχεία μας λέει ο κ. Γκάους. Είπατε επίσης ότι κατά τη δική σας άποψη να υπάρξει η εφαρμογή της ε, οδηγίας αυτής για τα συστήματα αυτά και αναφέρθηκε η γνωμοδότηση του Υπουργείου για το Opel Zafira ότι δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας των κινητήρων. Πώς έφτασε λοιπόν ε, πώς μπόρεσαν κάποιοι να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αρκούσε να υπάρξει μια αλλαγή των παραμέτρων του λογισμικού και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στα αποτελέσματα που είδαμε. Φυσικά μπορεί κανείς να επιτύχει καθαρότερα τους κινητήρες με τεχνικά μέσα. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν υψηλότερε ε, εκπομπές. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα και με μια χρήση λογισμικού. Το λογισμικό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί σε κάθε κινητήρα και σε κάθε, και κάθε αυτοκίνητο. Αυτά τα οποία έχουμε δει με τον κινητήρα diesel των 2 ε, λίτρων, ότι εκεί πέρα το software θα μπορούσε να έχει παίξει αυτό το ρόλο, αλλά για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, δεν ξέρουμε αν αυτό θα μπορούσε να είναι η, η απάντηση στις αποκλήσεις που έχουμε δει. Εμείς ε, επομένως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση του Ευρωπαϊκού Κύκλου Ελέγχου του ΕΝΕΔΕΤΣΕ. Ένα περαιτέρω ερώτημα. Είπατε στις ε, πρώτες σας απαντήσεις ότι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται χωρίς να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό. Αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να είχατε εσείς πρόσβαση στο λογισμικό, τι ακριβώς θα κάνατε. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας χωρίς να έχουμε τους απαραίτητους τους εμπειρογνώμονες για το λογισμικό. Δεν είναι όμως ο δικός μας σκοπός. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τέτοιες έρευνες Αυτό είναι θέμα των οργανώσεων καταναλωτών. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο από αυτό που κάνουμε. Εμείς βλέπουμε το όχημα ως ένα μαύρο κουτί και καταμετρούμε τις εκπομπές του και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι σε καλό επίπεδο και σε κακό επίπεδο. Η έρευνα για τα αίτια όλων αυτών των προβλημάτων θα πρέπει να γίνει από κάποιον άλλον, κατά πάσα πιθανότητα, από τον κατασκευαστή και τις επόσημες αρχές. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κύριο Σούτσο. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε μια συζήτηση με την ε, Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εμείς ε, ήμασταν κάπως επικριτικοί για αυτούς και τη στάση που έχουν κρατήσει. Ο κύριος Μπόκερ στις 16 Ιουνίου μας είπε από το Κέντρο για Ηλεκτρονική και Κινητήρες ε, καύσης μας είπε κάτι ενδιαφέρον. Και λέει ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση με, το, ε, με τον, τις μετρήσεις των κινητήρων, ότι κανείς δεν ασχολείται με τις πραγματικές ε, τιμές και αυτό είναι και μια πρόσκληση προς παραβάσεις όταν είναι ασαφείς οι, οι οδηγίες για την... Ε, ναι, η δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιούνται μηχανισμοί προστασίας του κινητήρα, ε, λέει ο κύριος Γκάους, αυτό οδηγεί σε μία ασάφεια. Υπάρχουν ε, ακραίες ίσως συνθήκες σε σχέση με την προστασία του, κινητήρα. Εμείς όμως δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μήπως τότε ο νομοθέτης δεν έχει ε, κάνει συγκεκριμένη τη θέλησή του, οπότε η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά της ε, την νομοθεσία. Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίηση, θα πρέπει να αναφέρονται με σαφείς τρόπους οι ομαλές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα και επομένως θα πρέπει να γίνεται και σε ε, συγκεκριμένες θερμοκρασία θερμοκρασίας και να αναφέρονται σαφώς. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι οι αρχές ερμηνεύουν διαφορετικά αυτό τον, ε, αυτή την ε, οδηγία. Δεν μπορώ παρά μόνο εικασίες να εκφράσω. Φυσικά τα διαφορετικά κράτη μπορεί να έχουν διαφορετικά εργαστήρια και διαφορετικές αρχές που κάνουν τον έλεγχο. Προφανώς <clears throat> θα ήταν ευχής έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την ε, εφαρμογή αυτών των ε, προδιαγραφών. Και τα εργαστήρια δεν πρέπει να λειτουργούν λες και πέσουν στην ε, αγορά και πρέπει να έχουν καλούς πελάτες. Ε, Μήπως θέλετε εσείς να εξασφαλίσετε ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να μειώσουν την, ε, ε τις εκπομπές των οχημάτων και οι καταναλωτές θα έπρεπε να πληροφορηθούν ότι είναι σημαντικό να, παίζουν, να ελέγχουν περισσότερο την ποιότητα των εκπομπών. Φυσικά, με χάρη στην ε, δημοσιότητα που δόθηκε στα μέσα ε, ενημέρωσης, οι, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο και για την ασφαλειά τους, αλλά και για την, τις εκπομπές των καυσαέριων. Ο κύριος Έρτουγκ. Εγώ επανέρχομαι στο ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος από τους Πρασίνους, ο οποίος έθεσε το ερώτημα για το πότε δώσετε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για τις αποκλήσεις από τις ε, οριακές ε, ε, αρχέ, ε, τιμές που ε, μετρήθηκαν. Τα δώσατε αυτά τα στοιχεία ή όχι. Εμείς μόνο όταν βλέπουμε διαφορετικές, μεγάλες διαφορές από τον ευρωπαϊκό κύκλο, το NDC, τότε δίνουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Αν τώρα είμαι εκτός από την, έξω από τη αυτό μόνο στη διαδικασία έγκρισης τύπου, εάν υπάρχει ε, μια τέτοια ε, περίπτωση εκτός τύπου, εκτός τύπου δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπήρξε σε αυτήν την περίπτωση κάποια ε, πληροφόρηση των αρμοδιών υπηρεσιών, λέει ο κύριος Ερτούκ. Έχει γίνει κάτι τέτοιο τους τελευταίους μήνες, παραγωγός Και επίσης, ε, ποια είναι η θέση σας για το ECOTEST. τα αυτοκίνητα αυτά που ανέφερα στις ε, διαφάνειες, όλα αυτά τα οχήματα πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα την ένδυση τύπου. Αλλά βλέπετε μετά με τον παγκόσμιο κύκλο, το ΔΕΛΤΕΣΕ, ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως η αρμόδια αρχή όταν υπάρχουν υψηλές εκπομπές εκτός του κύκλου δοκιμασιών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση νομική να αναφερθεί αυτό. Και τα στοιχεία αυτά για, την, ε, για, τον, ε, για το οικολογικό τεστ είναι πράγματα όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται ή όχι. Φυσικά υπάρχουν τα μεσαία ενημέρωση τα οποία ενδιαφέρονται. Είχαμε περιπτώσεις όπου υπήρξαν υψηλές τιμές για οξύδια του ασότου ή και για σωματίδια. Φυσικά. Δεν έχει γίνει κάτι επισήμω συγκεκριμένο. Φυσικά τώρα η κοινή γνώμη ε, στη Γερμανία έχει εντυπωσιαστεί, έχει ε, ουσιαστικά ευαισθητοποιηθεί περισσότερο από την ε, απόφαση που ελήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Βυζίκη. Ευχαριστώ κύριε Γκάουσου. Ε, δεύτερο... Ευχαριστώ Ποια είναι η σχέση... Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε τι, οικονομική ενδεχομένως σχέση βρίσκεται η ΑΝΤΑΚ με τις αρμόδιες αρχές. Για τα θέματα των εκπομπών, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση ε, επιχειρηματικού τύπου με ε, εταιρείε ή με κάποιον άλλο. Εμείς έχουμε μια απόλυτη ανεξαρτησία στα θέματα αυτά και φυσικά μπορούμε να πάρουμε ε, να μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι, κάτι τέτοιο για τα θέματα αυτά. Η πρακτική λοιπόν αυτή που έχετε που έχετε τα 150 οχήματα που δοκιμάζετε το χρόνο. Εσείς πώς διαλέγετε αυτά τα οχήματα, τα, τα αγοράζετε, τα μισθώνετε, τι κάνετε. Είναι συνήθως ε, οχήματα που δίνει ο κατασκευαστής, τα οποία τα χρησιμοποιούν, για ε, δοκιμασίες από τα περιοδικά των αυτοκίνητων παραγωγής χάρη είναι αυτοκίνητα του κατασκευαστή. Δεν έχουμε άλλο εναλλακτικό τρόπο να ελέγξουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα Επίσης θα δοκιμάσουμε, δίνουμε τις πληροφορίες και στον ε, κατασκευαστή για τα αποτελέσματα των ε, δοκιμασιών και μετά τα αποτελέσματα αυτά ε, δημοσιεύονται και ενδεχομένω με κάποιο σχόλιο του κατασκευαστή. Άμα δείτε έντυπα από στο Motorvert, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές φορές τα σχόλια του κατασκευαστή. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις δοκιμές εκπομπών που πραγματοποίησατε, τι ποσοστό οχημάτων σέβεται τα όρια, τηρεί τα όρια, ποιο το ποσοστό οχημάτων που ξεπερνούν μια μισή φορά το όριο και τι ποσοστό οχημάτων ξεπερνούν πάνω από 2% σε σχέση με το δίκτυο συμμόρφωσης. Πιστεύετε εξάλλου ότι η επιλογή αυτή του 2.1 και 1,5 τεχνολογικά δικαιολογείται. Ευχαριστούμε. Μέχρι τώρα πρέπει να σας πω ότι οι δοκιμές RD ε, δεν έχουν ε, γίνει, δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα τέτοιο βαθμό που να μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες ενδείξεις. Έχουμε κάποια βάση Πρόκειται για ένα, μια δοκιμή πραγματικού κύκλου για το διοξίδιο του άνθρακα και αυτό αποτελεί τη βάση που χρησιμοποιούμε και για το real world emission. Δεν μπορώ να σας πω λοιπόν ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσοστό για το 2,1 ή 1,5 ή 2. Έχετε την μπλε κολόνα και μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποια οχήματα μπορεί να είναι εντάξει, αλλά οι τρεις δοκιμές RDE που κάναμε δεν ε, έδειξε κανένα αυτοκίνητο να πετυχαίνει 100%. Όσον αφορά τις απόλυτες τιμές, απαιτούμε 1,5 δίκτυ. Δεν θεωρούμε ότι πόσο να θα πρέπει να βάλουμε το 1,1. 1,5 είναι καλύτερο από το τίποτα. Αν αυτό αποτύχανε, τότε θα ήταν καταστροφή. Το 1,1 και 1,5 τεχνικά μιλώντας και όσον αφορά το κόστος δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Είναι ένα περιθώριο ε, ελιγμών που επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Σίγουρα, όσο περνά ο καιρός, θα έχουμε όλο και περισσότερα οχήματα τα οποία θα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή που θα τηρούν το 1,5. Είχα δύο φορές χρόνο ομιλίας, οπότε θα το χρησιμοποιήσω μια και έξω, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε. Στο έγγραφο του 2015 λέγατε ότι οι τελευταίες τεχνολογίες σέβονται τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές απόλυτα. Πόσα οχήματα τηρούν όντως τις προδιαγραφές αυτές και γιατί δεν είναι περισσότερα. Απάντηση. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα απόλυτα αυτό το οποίο με ρωτάτε. Ε, σε ποιο έγγραφο αναφέρεστε ακριβώς? Position Paper της ADAC που είναι το 2015. 70 του 2015. Για ντίζελ. Δεν έχω όλο τον τίτλο, λέει η κυρία Ρεβό. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Τα Okay. And wir sagen, Η τεχνολογία υπάρχει για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η ανακύκλωση των καυσεαρίων και το σύστημα HR Η τεχνολογία αυτή άμα χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Και αυτό το έχουμε πει ήδη. Και έχουν ζητήσει να χρησιμοποιηθεί ένας παράγον διόρθωσης 1,5 γιατί αυτό θεωρούσαμε ότι ήταν εφικτό. Το υπόλοιπο το κομμάτι τη δεν, πα, δεν παρακολούθησα ακριβώ τι ερούσατε. Όχι, εγώ θέλω να ήξερα το ποσοστό των οχημάτων που ήδη από τώρα συμμορφώνεται. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες. Η κάθε τεχνολογία έχει τα στοιχεία που μπορούν να επιτύχουν το στόχο αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ένα όχημα το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει με παράγοντα συμμόρφωση 1,5 στις πραγματικές συνθήκες τις προδιαγραφές αυτές. Όσα, αν υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα θα πρέπει να υπάρχουν λίγα, αλλά για μας είναι απόλυτα εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, γραπτά ίσως καλύτερα. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Ντάλτον. Κύριε Ντάλτον. <laughs> Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ο κύριος Δεμασμάκερ νομίζω έχει ζητήσει το λόγο. Ωραία. Ευχαριστώ. Α, ούτε εσείς, όχι. Καλώς. Παρακαλώ λέει ο κύριος Ροσόλ. Ευχαριστώ κύριε Ντάλτον που μου δίνετε τη σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Γκάους, εσείς εδώ εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των οδηγών. Πιστεύετε ότι οι οδηγοί υπογόρασαν οχήματα τα οποία τελικά ρηπαίνουν περισσότερο από όσο προβλεπόταν θα έπρεπε να πάρουν αποζημιώσεις. Η The Welt, η γερμανική, αλλά όχι και μόνο αυτή η εφημερίδα και άλλες είπαν ότι 5.000 δολάρια πρέπει να δώσει σε καθένα από τους οδηγούς ε, Volkswagen Diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν για τους Γερμανούς καταναλωτές και η δικιά σας η οργάνωση, λες, και τι σκοπεύει να κάνει από αυτού. Τι νομίζει, ποια είναι η γνώμη της. Αυτή είναι μια πολιτική ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ σε εμπειρογνώμων να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Εμείς προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της τροποποίησης των κινητήρων στην Volkswagen που οδηγούν σε μεγαλύτερο κόστος ε, καυσίμων. Προφανώς μπορεί να διεκδικήσει κανείς το πρόσθετο κόστος το οποίο προκύπτει αλλά τώρα για μια καταποκοπή αποζημίωση για το καταναλωτή αν ε, έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τα προβλήματα αυτά που έχουν ε, ε αναφερθεί. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ ως ε, τεχνικός. Ο κύριος Ροσφόρ. Ωραία. Σαν μηχανικός θα ρωτήσω. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι το Volkswagen με την χρήση του λογισμικού που παρακάμπτει θα είχε μεγαλύτερη αξία αν δεν είχε γίνει αυτή η απάτη. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, πέρυσι πουλήθηκαν λιγότερα Volkswagen ως μεταχειρισμένα, έτσι δεν λέω ως καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα. Δηλαδή υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι δυσκολεύτηκαν ή ανέβαλαν την ε, διάθεση στην αγορά των δικών του οχημάτων για να τα πουλήσουν σαν μεταχειρισμένα. Εσεί, σαν μηχανικό, λοιπόν, πιστεύετε ότι ο ιδιοκτήτη ε, ενό οχήματο Volkswagen στη Γερμανία, στην Ευρώπη γενικά σήμερα έχει στα χέρια του ένα αγαθό που αξίζει λιγότερα από όσο θα ήταν αν δεν είχε αυτό το λογισμικό και δεν θα ήταν φυσιολογικό να αποζημιωθεί. Δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως και ο Αμερικανός καταναλωτής, γιατί στην Αμερική το έχει αποδειχτεί η ίδια η Volkswagen να δώσει την αποζημίωση. Απάντηση η Volkswagen κάνει αυτήν την ε, τροποποίηση του οχήματος ώστε το αυτοκίνητο να μην είναι χειρότερο από ότι πριν από αυτή την αλλαγή, δεν μπορώ να πω ότι, το, ότι πρέπει να υπάρξει αποζημίωση. Αν η Volkswagen μπορεί να επαναφέρει το όχημα στην κατάσταση που ήταν στην αρχή, χωρίς να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και μειώσεις στην απόδοση του οχήματος, στην περίπτωση αυτή δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη μια αλλαγή. Αυτό μπορώ να σας το πω. Γι' αυτό έχουν γίνει και οι ανακλήσεις ε, ορισμένων οχημάτων. Σούτσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και το άκουσα αυτό ότι στη Γαλλία έχουν πέσει ορισμένα αυτοκίνητα σε τιμή μεταπόληση. αλλά επί, της, ε, επί του θέματο και πάλι υπάρχουν πολλέ ε, δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει για την θέση των πολιτών, γιατί ε, διαλέγουν τα αυτοκίνητα επειδή είναι πιο δυνατά ή επειδή είναι πιο φτηνά σε καύσιμο. Έχετε κάνει εσείς κάποιες δημοσκοπήσεις μεταξύ των πελατών σας ή μεταξύ των, των μελών σας για τα θέματα αυτά. Δεν ε, έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά το θέμα της, των εκπομπών είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει τους καταναλωτές πολύ λιγότερο από το θέμα της ασφάλειας. Ακόμα και για τα θέματα της ασφάλειας ο καταναλωτής δεν είναι έτοιμος να δώσει πολύ περισσότερα. Παραδείγματος χάρη ένα σύστημα υποβοήθηση της οδήγησης ε, δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση αυτοκινήτων. Και υπάρχουν και... Δεν μπορώ να σας πω τώρα τι γίνεται με τα άλλα εξατήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις εκπομπές ή την ασφάλεια των οχημάτων. Ένα άλλο ερώτημα. Για το τεστ σύγκρουσης. Έχουμε δει ότι οι κατασκευαστές έχουν προσαρμόσει ουσιαστικά τα οχήματά της για τις δοκιμασίες εκπομπών. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει γίνει κάτι αντίστοιχο για τα τεστ σύγκρουσης, ότι έχουν προσαρμοστεί τα αυτοκίνητα να αντέχουν σε αυτά τα συγκεκριμένα τεστ και μόνο. Έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο στα crash test, τα τεστ σύγκρουσης και έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο Έχουμε πολλές ε, συζητήσεις έχουν γίνει για να δούμε όλα τα, τα πράγματα τα οποία μπορούν να δοκιμαστούν στα πλαίσια των συγκρούσεων. Και υπάρχει πάντα μια ομάδα ε, εργασίας η οποία εξετάζει τα θέματα αυτά και επομένως ε, προηγούνται, προπορεύονται τις νομοθεσίες. Υπάρχουν τα συστήματα αυτά για αυτόματη πέδηση, για το να λειτουργούν οι ζώνες ασφαλείας εκ των προτέρων κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν εξασφαλιστεί, κυρία Κιωστινιά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα ίσω. Είχαμε δει στην προηγούμενη μας ακρόαση παραδείγματα ότι η εγκινήσει ε, οι δοκιμές εγκινήσει δεν είχαν δώσει ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσματα. Ήταν ασαφή τα αποτελέσματα. Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτά. Μπορώ να σας πω ότι δεν πρόκειται να ακυρωθεί η μέτρηση στο εργαστήριο με τη χρήση των εγκινήσει, των κινητών μετρήσεων. Αλλά πρέπει να υπάρξει, υπάρχει ο φόβος ότι οχήματα τα οποία έχουν καλή απόδοση στις εργαστηριακές ε, δοκιμασίες δεν έχουν την αντίστοιχη συμπεριφορά στον δρόμο. Αυτό, γι' αυτό πρέπει εμείς να έχουμε και δοκιμασίες στον δρόμο. Αλλά μόνο δοκιμασίες στον δρόμο δεν είναι η σωστή λύση. Μπορείτε όμως να πείτε αν κατά την άποψή σας κάποτε η τεχνολογία μέτρηση σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο. Εμείς δεν, δεν έχουμε εμπλοκή στην ε, ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά έχουμε κάνει τις πρώτες δοκιμές με κινητές μονάδες μέτρησης και έχουμε και επαφή με αυτούς οι οποίοι παράγουν τις συσκευές για κινητή ε, δοκιμασία εκπομπών και μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις όπως κάνουν και οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ε, ελέγχου των, ε, το, τον Μπορούμε έτσι με τον τρόπο αυτό να βελτιώσουμε την τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία είναι σχετικά νεοφανής. Και είναι πάρα πολύ σωστό να ανταλλάγουμε πληροφορίε. Εμείς βέβαια δεν εμπλεκόμαστε στην έρευνα για τη βελτίωση αυτών των τεχνικών. Δεν έχετε λοιπόν πρωτοβουλίες αυτές αλλά μπορείτε, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η τολή τεχνική που χρησιμοποιείτε, μπορείτε εσείς ε, να εκφράσετε κάποια άποψη για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι αναξιόπιστες ακόμα απόλυτα αυτές οι, οι μετρήσεις στο δρόμο, απλώς υπάρχουν, επηρεάζονται από πολλά πράγματα, από, την, από τον άνεμο, παραδείγματος χάρη μπορεί να επηρεαστούν, από τη διαφορά της ε, θερμοκρασίας, από διαφορετικές συνδίκες θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης και φυσικά όταν μετράει κανείς κάτι σε συνθήκες βροχής μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά διαταράσσουν λοιπόν την ε, μέτρηση. Αλλά σας λέω και πάλι δεν θα γίνουν ποτέ οι εργαστηριακές ε, δοκιμασίες περιπές. Επανέρχομαι στις πραγματικές συνθήκες λέει ο κύριος Ερτούκ αν έχουμε μια επαρκή και πλήρη διαδικασία δοκιμασίας σε πραγματικές συνθήκες, αυτό μπορεί να αποκλείσει την ε, απάτη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την αποκλείσει απόλυτα, απλώς θα έχουμε καλύτερες συνθήκες για να το διακριβώσουμε. Ο στόχος μας, όπως και με τις οικολογικές ε, ε δοκιμασίες, Νομίζω ότι ενδεχομένω θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερη δυνατότητα πληροφορι... περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο δοκιμασιών. Αν είναι καλές δοκιμασίες θα έχουμε πολύ καλύτερη γνώση. Και δεν σας ενδιαφέρει να εξετάσετε τις ε, στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές για να παραπλανούν τις δοκιμασίε. δοκιμασίες. Μα εδώ όταν δοκιμάζει κανείς και με, ε, σε, σε χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει και εκεί να υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση. Ενδεχομένως ε, οι στρατηγικές, άμα, άμα ελέγχουμε σε πολλές θερμοκρασίες, τότε οι τεχνολογίες παραπλάνησης μπορεί να λειτουργούν μονάχα σε ακραίες συνθήκες. Τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι πληροφόρησατε την Ομοσπονδιακή Αρχή για τα οχήματα ότι το αντάτς βρήκε κάποιες αποκλήσεις από τις τιμές. Έχει γίνει αυτό πριν από το 2012 και έχετε δει αυτή την αλλαγή σε, στους, στη μέτρηση NDC μεταξύ ε, ψυχρής, ψυχρών συνδικών και θερμών συνδικών. Δεν ξέρει όμως η Ομοσπονδιακή Αρχή πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Οι αποκλήσεις είναι κάτι που αφορούν τις αρχές και ο... δεν υπάρχει <clears throat> ε, ένα νομικό πλαίσιο ώστε να κάνει κάτι κανείς εφόσον δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για τα θέματα αυτά. Είναι κάτι λοιπόν όμως αυτό το οποίο το έχουν αποφασίσει οι αρχές ότι ό,τι γίνεται εκτός του κύκλου δοκιμασιών δεν έχει καμία σημασία σε νομικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ε, εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ επίσημα κάποια καταγγελία αυτού του είδους. Και οι αρχές λένε ότι εφόσον στο επίπεδο του ένεται τα πράγματα γίνονται καλά, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Όχι, δεν είπανε ποτέ κάτι τέτοιο. Και υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση, γιατί όταν είναι ε, σε θερμές συνθήκες ε, στον κύκλο σε πρέπει να είναι μεγαλύτερες οι εκπομπές, μα όταν υπάρχει σε υψηλότερη ε, θερμοκρασία ο κινητήρας, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή οξυδίων του αζότου. Και άμα είναι ψυχρός ο κινητήρας είναι λιγότερες οι παραγωγές ε, οξυδίων. Αλλά δεν βλέπω κάποιο λόγο να γίνεται αυτό εάν είναι καλά κατασκευασμένοι το τεστ. Εσείς λέτε ότι ένας παράγων συμμόρφωσης 1,5 είναι εφικτός. Αυτό το βασίζεται στις μετρήσεις που έχετε κάνει. Πόσο μεγάλες είναι οι αποκλήσει αν χρησιμοποιήσει κανείς το τεστ των ε, ελαφρών οχημάτων, το παγκόσμιο τεστ ε, ελαφρών οχημάτων και το συγκρίνει με το, τις μετρήσεις των δρόμων. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια μέτρηση που να δείξει το 1,5 αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τεχνικά ε, εφικτό και αυτό μπορεί να αφορά και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Μα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει ο παράγων ε, ε συμμόρφωσης να βοηθά τους, κατα... τους κατασκευαστές για να πιάνουν τις προδιαγραφές, απλώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει μονάχα για να καλύπτει το σφάλμα μέτρησης. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο τμήμα αυτό της ακρόασης. Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και όπως είπα θα σταλούν και γραπτά κάποιες ερωτήσεις ε, από μας προς εσάς. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας μέχρι τώρα. Um, Παρακαλώ τώρα τον κύριο Νίκ Μόλτεν να έρθει εδώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίκ Μόλντον. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Η Emission Analytics είναι μία εταιρεία ανεξάρτητη που κάνει δοκιμές. Έχουμε συζητήσει πολύ γι' αυτό ε, κάνει μετρήσεις όσον αφορά την ε, πραγματική, σε πραγματική κατάσταση, ε, σε συνθήκες οδήγησης δηλαδή. Εν μία ώρα και 40 λεπτά θα κρατήσει εδώ η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας, αλλά στην αρχή έχετε 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω ποιοι είμαστε. Είμαστε σχετικά νέοι στον χώρο. Έχουμε τρεις συγκεκριμένους τομείς τους οποίους δραστηριοποιούμεθα για τα δεδομένα και τις δοκιμές τις οποίες κάνουμε. Ε, έχουμε ιδρυθεί εδώ και πέντε χρόνια, ίδρυσα αυτήν την ομάδα για έναν λόγο, να παρακολουθήσουμε και να έχουμε εκθέσεις από πλευράς των καταναλωτών σε σχέση με τις διαφορές τις οποίες έβλεπαν στην πραγματική τους κατανάλωση σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγαν τα εγχειρίδια χρήση και οι διαφημίσεις των αυτοκινήτων τους. Αυτό μου προκάλεσε ενδιαφέρον, γιατί εγώ ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες αποκλήσεις και αποφασίσαμε λοιπόν να το διερευνήσουμε το θέμα και να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο, όπως και ο νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Δοκιμών και το πρωτόκολλο των ελέγχων των δοκιμών γύρω από αυτό. Τώρα, προσπαθήσαμε λοιπόν εμείς να δούμε αν μπορούμε να δούμε τα πράγματα καλύτερα. Μετά από πολλές έρευνες αποφασίσαμε ότι είναι δυνατόν μέσω της χρήσης των λεγόμενων φορητών συστημάτων μέτρησης και της ανάλυσης των δεδομένων να μπορέσουμε να έχουμε εναλλακτικά συστήματα στην διάθεσή μας. Το πετύχαμε αυτό, συλλέξαμε κάποια χρήματα, επενδύσαμε ε, σε εξοπλισμούς TEMS, χρησιμοποιήσαμε επίσης ε, και ε, μηχανολόγους και αρχίσαμε να κάνουμε δοκιμές στα αυτοκίνητα. Έχουμε ελέγξει μέχρι τώρα πάνω από 1.200 αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε άλλες χώρες και στη ΣΥΠΑ. Και εγώ σήμερα αυτό που σας παρουσιάζω είναι ο καρπός των δοκιμών PEMS που κάναμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω κρίση σε επίπεδο εκπομπών στο μέλλον. Έχει σημασία για μένα να πω ότι για μας η μελέτη αυτή δεν ήταν άπαξ ενδιαφέρουσα. Το θέμα είναι να μπορεί να το κάνει κανείς με ένα κυλιόμενο τρόπο, έτσι ώστε να ελέγχει τα αυτοκίνητα τη στιγμή που τίθεται σε κυκλοφορία. Έχουμε τρεις βάσεις, στην Στουτχάρδη και στο Λος Άντελες. Έχουμε ελέγξει πάνω από 500 αυτοκίνητα, έχουμε δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές για επιβατηγά, αν και κάνουμε βέβαια και εμπορικά, εμπορικής χρήσης, δημόσιας χρήσης και φορτηγά και ε, διαθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε όλους τους εμπλεκομένους στην αγορά, δηλαδή καταναλωτές, κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, κατασκευαστές, εμπόρους κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν βλέπω το πράγμα αυτό, εγώ δεν είμαι μηχανολόγος, εγώ είμαι οικονομολόγος και θεωρώ εδώ ότι έχουμε μία αποτυχία της αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αφορά μια δυσλειτουργία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι καταναλωτές όταν έχουν να επιλέξουν έχουν μια τεράστια γκάμα αυτοκινήτων και τους δίδονται ε, πληροφορίες οι οποίες στην ουσία παραπληροφορούν και σε σχέση με τα νόξ, το άζωτο δηλαδή, και σε σχέση με το μέγεθος, το ύψος της κατανάλωσης και αυτό οδηγεί τους πολίτες να αγοράζουν το λάθος αυτοκίνητο. Μιλάμε για μια αποτυχία της αγοράς και πρέπει επιτέλους να διορθωθεί. Αυτά είναι τα καθημερινά μας κίνητρα. Λοιπόν, αυτά για το παρελθόν μας. Τώρα, ε, τρεις τομείς θα ήθελα να δω. Αυτό που μας επιτρέπουν να κάνουμε τα δεδομένα μας. Πρώτον, να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που ακολουθείται. Σας δώσω κάποια στοιχεία μόνο. Πρώτον, να δούμε το κενό ανάμεσα στις πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και στις επίσημες μετρήσεις. Και αυτό αφορά και στην κατανάλωση καυσίμων. Αυτό το οποίο βρήκαμε και δεν εκπλήσει κανένας είναι ότι οι πραγματικές εκπομπές είναι ψηλότερες από τις επίσημες. Αλλά για τη βενζίνη δεν αυξάνεται η διαφορά, αλλά αυξάνεται για τα πετρελαιοκίνητα. Βλέπετε με πορτοκαλί την γραμμή ε, των πετρελαιοκινητήρων, ενώ οι βενζινοκινητήρες είναι με μπλε. Αν δούμε επίσης ε, και ε, χρονικά το θέμα, υπάρχει μία άποψη ότι συνεχώς μειώνουμε την κατανάλωση και όλα πάνε καλά. Όχι βέβαια, Υπήρξε μια ουσιαστική τέτοια τάση μακροπρόθεσμη, αλλά από τον προηγούμενο χρόνο για πρώτη φορά υπάρχει αναστροφή. Οι επίσημοι αριθμοί δίδουν μια ψευδέστηση προόδου σε σχέση με το ύψος της κατανάλωσης. Οι πραγματικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξάνονται δυστυχώς και ιστορικά οι μειώσει ήσαν μικρότερε από ό,τι μα οδηγούσαν να πιστεύουμε οι επίσημοι αριθμοί. Αυτό ισχύει και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη. Δεν έχουμε μόνο ένα θέμα λοιπόν με τα νόξα, αλλά έχουμε θέμα επίσης και με τα διοξίδιο, το διοξίδιο του άνθρακα. Ένας άλλος τρόπος είναι να συγκρίνουμε τα δεδομένα ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ευρωπαϊκές δοκιμές και τις αμερικανικές δοκιμές γιατί υποτίθεται ότι σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα είμαστε μακράν μπροστά. Όχι βέβαια. Αυτό το οποίο σας δείχνουμε εδώ είναι η κατανάλωση ε, βενζίνης η οποία συγκλίνει με την ε, ευρωπαϊκή βενζίνη και τους κινητήρες τους βενζινοκίνητους και τις εκπομπές σε διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό οφείλεται στους πολύ αυστηρούς στόχους που επιβάλλει στην αυτοκινητοβιομηχανία επιβατηγών η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν έχουμε ηγέτιδα θέση σαν Ευρώπη, αλλά συνολικά για το σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων είμαστε ε, υψηλότερα, ιδιαίτερα σε σχέση με το πετρέλαιο. Και γι' αυτό ε, βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είναι αυτό το οποίο μας δίδει το πλεονέκτημα σε σχέση με την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, το θέμα είναι αν υπάρχει δυνατότητα αντισταθμίσεων ανάμεσα στο διοξίδιο του άνθρακα και στις εκπομπές οξυδίου του αζότου, δηλαδή αν η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα είναι το τίμημα της μείωσης του νόξου. Δεν υπάρχουν αποδείξεις απόλυτες, αλλά υπάρχουν κάποιες τάσεις οι οποίες για πρώτη φορά δείχνουν ότι εμείς είχαμε ε, παρακολουθήσει με την μπλε γραμμή την κατανάλωση. Για πρώτη φορά είδαμε ότι το 2015 έπεσε η κατανάλωση καυσίμων για πρώτη φορά. Αυτό ήταν μια εποχή επίσης πίεσης και συγκέντρωσης της προσοχής και υπογράμμισης του οξυδίου του αζότου και νομίζω ότι ο ανταγωνισμός αυτός σε σχέση με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων είναι κάτι το οποίο πράγματι ισχύει και υπάρχουν και τεχνικά θέματα σε σχέση με το τίμημα όπως η χρήση του EGR και των καθαρών παγίδων ή συστημάτων παγίδευσης NOx. Ελέγξαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα εδώ και πολλά χρόνια και βλέπουμε ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες τάσεις. Νομίζω ότι εδώ βλέπουμε και τους παράγοντες συμβατότητας, τους παράγοντες συμμόρφωσης σε σχέση με τα αυτοκίνητα που ελέγξαμε. Η μπλε γραμμή είναι ο μέσος όρος των 12 μηνών. Εμείς ε, κολλήσαμε στα Europe 5, στα ε, ε, ε, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι τα προβλεπόμενα. Υπήρξαν βελτιώσεις το 2014 που τέθηκε σε κανονισμό το Euro 6 το οποίο στην ουσία με συνδυασμό, σε συνδυασμό με την απειλή των νέων κύκλων δοκιμών οδήγησε στη μείωση του νόξ. Αλλά μετά από μία περίοδο, αν θέλετε, έξι μηνών βελτίωσης, τα πράγματα μετά κόλλησαν και δεν είδαμε από εκεί και πέρα μείωση σε πραγματικούς αριθμούς των νόξ και είμαστε πάντα τέσσερις φορές παραπάνω για τα νέα οχήματα. Δεν θα επιμείνω σε αυτό αλλά βλέπετε εδώ μια κατανομή των δεδομένων ανάμεσα στο SCR και στα LNT, στις δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Τα SCR λέγεται ότι είναι καλύτερη τεχνολογία από τα LNT και αυτό δεν είναι αλήθεια τεχνολογικά, γιατί υπάρχουν αναπτύξεις LNT σωστές και καλές και SCR αναπτύξεις κακές. Και τέλος τα νέα αντί θα βοηθήσουν οι νέες πραγματικές συνθήκες δηλαδή δοκιμών. Το θέμα είναι ότι το 30% των Euro 6 που είναι στην αγορά θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου συμβατότητας συμμόρφωση. Δηλαδή αυτό το 2,1 δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρό δεν πρέπει να αλλάξουν και πολλά σε επίπεδο, αν θέλετε, μηχανισμών για να το πετύχουμε. Το RDE θα είναι αποτελεσματικό όταν πέσουμε στο ποσοστό συμμόρφωσης 1,5 και κάτω από το 1,5. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξουν αλλαγές πολλές. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Τα δεδομένα που συλλάγουμε είναι διαθέσιμα με συνδρομές. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Εμείς δεν ε, ε, δημοσιεύουμε μόνο τους τίτλους των εργασιών μας, το σύνολο των στοιχείων και των δεδομένων είναι στη διάθεσή σας. Χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα για να φτάσω, να ξανά στους καταναλωτές. Έχουμε περάσει στην δημοσίευση του λεγόμενου δίκτυ ποιότητας του αέρα Equa είναι στην ουσία μια διαδικασία που διακρίνει αν θέλετε τις καταστάσεις, δεν είναι θα έλεγα μια νομική ρύθμιση, έχει οκτώ βαθμίδες, το α είναι το, το A αγγλικό είναι το καθαρότερο και το H αυτό που μολύνει περισσότερο. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Από το α μέχρι το γ όμως έχουμε πετύχει τον δείκτη συμμόρφωσης 2,1 είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μας σε σχέση με το πρόγραμμα Equa και νομίζω είναι ότι όλα τα πετρελαιοκίνητα Euro 6 μόνον 7 έχουν πάρει A και μόνο ένα από αυτά είναι από την ομάδα από βιομηχανιών Volkswagen, τον όμιλο Volkswagen. Αυτό δεν αφορά, επαναλαμβάνω, ε, τα, ε, τα, τους τελευταίους τύπους Euro 6 αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ε, ε, κάποια στοιχεία, θα έλεγα μη προφανή, ε, τα κάποια μαθήματα τα οποία μπορεί να βγάλει κανείς, κάποια συμπεράσματα από όλες αυτές τις διαβαθμίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόλτεν. Οι εισηγητές μας πρώτα, κύριος Γεβραντή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόλτεν, για την παρουσίασή σας. Για μας, ο κύριος λόγος για την έρευνα αυτή που κάνουμε εδώ είναι να δούμε αν και γιατί κάτι δεν πάει καλά και αν υπήρξε κάποια κάλυψη, ένα σκέπασμα από τις δημόσιες αρχές. Και εσείς ε, πολύ καλά λέτε γιατί ξεκινήσατε με την ε, εταιρεία σας, γιατί σας έκαναν εντύπωση διαφορές ε, που υπήρχαν στις δοκιμές που γινόντουσαν στα εργαστήρια και εκείνες που γινόντουσαν σε πραγματικές συνθήκες. Οπότε και για τα οξύδια του ζώτου, Το γενικό ερώτημα είναι, μας ξεγέλασε η αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να αισθανόμαστε ότι οι δημόσιες αρχές κουκούλωσαν τα πράγματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσει κανείς είναι η εμπειρία που έχω για όλη την διαδικασία. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ σαν κάποια ισχυρή οργάνωση όπου οι κυβερνήσεις θα μας ακούσουν κτλ. Εμείς ξεκινάμε, έχουμε ως αφετηρία το ότι είμαστε μια startup ε, βρετανική εταιρεία και προσπαθούμε να ακουστεί η φωνή μας. Και πώς το κάναμε αυτό. Πρώτα απ' όλα δημοσιοποιώντας τα αποτελέσματα των δοκιμών μας για την κατανάλωση καυσίμων, τελευταία το 2014 και όλη αυτή την περίοδο και εγώ συμμετείχα σε διάφορες διασκέψεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για να τους εξηγήσω ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, όπως κάνω και εδώ σήμερα. Αυτά από το 2012. Και οι διασκέψεις ε, αυτές ήταν με εκπροσώπους από διάφορες αρχές ρυθμιστικές, κυβερνητικούς εκπροσώπους, αλλά και εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή, όλο αυτό το καιρό, αυτό ακριβώ κάνουμε. Φροντίζουμε να ακουστεί η φωνή μα. Βέβαια, χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αρχίσει ο κόσμο να καταλαβαίνει ότι πράγματι διαθέτουμε στοιχεία τα οποία αξίζει τον κόπο να καθίσουν και να τα ακούσουν και ότι έχουν τη σημασία του. Οπότε η εμπειρία μου είναι ότι είναι δύσκολο για μένα να πω, κοιτάξτε, γράψαμε στην τάδε κυβέρνηση και είπαμε ότι γίνεται αυτό και αυτό. Και ξέρω ότι εκείνοι δεν αντέδρασαν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μας έχουν ακούσει. Έπειτα να ξέρετε ότι ακόμα και το ICCT όταν έκανε τη δικιά του αναφορά τα μισά στοιχεία ήταν από εμά. Τότε άρχισε η φωνή μας να ακούγεται. Οπότε υπάρχει κάποιο σημείο από το οποίο αρχίσαμε να ακουγόμαστε από το Ευρω 6 αν υπήρχε κουκούλωμα, όχι, δεν ξέρω, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε καμιά υποχρέωση κάποιος να μας εισακούσει. Ε, Γκεμπράντη, θέλω να έρθω σε μία φράση στις απαντήσεις σας. Μιλάτε για τον ε, ε, ευγενή τρόπο ε, δοκιμών του NEDC. Σαν να λέτε ότι είναι εύκολο τελικά να περάσει κανείς αυτή την δοκιμή και ότι δεν έχει τελικά και πολύ σχέση με την πραγματικότητα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο κύκλος δοκιμών έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο εύκολο για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συμμορφωθούν, δηλαδή να έχουμε πιο καθαρό αέρα στους δρόμους μας στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, ε, πριν από μας υπάρχει το NEDC και δεν νομίζω ότι φτιάχτηκε επίτηδες για να είναι μια εύκολη δοκιμή για να περνάνε εύκολα και να εγκρίνονται τα αυτοκίνητα. Ήταν για σύγκριση όσον αφορά ε, την κατανάλωση. Φτιάχτηκε με καλές προθέσεις, αλλά δεν ε, τροποποιήθηκε ποτέ. Δεν προσαρμόστηκε ποτέ στα προβλήματα τα οποία σιγά σιγά προέκυπταν και που ήταν η αποτυχία. Σε αντίθεση με την νομοθεσία στις ΗΠΑ, όπου είχαν αντίστοιχα προβλήματα με έναν κύκλο του FTP, δηλαδή που εφάρμοσαν εκεί, Συνεπώς θα έλεγα ότι απέτυχε η αποστολή μας. Ερώτηση και πιστεύετε ότι επίτηδες δεν προσαρμόστηκε. Γιατί το ότι είχε παλιώσει, ότι δεν ανταποκρινόταν σε απαιτήσει της πραγματικότητας, αυτό ήταν κάτι κατάφορο. Γιατί δεν προσαρμόστηκε. Επίτηδες. Απάντηση. Η άποψή μου είναι ότι ο κόσμος προτιμάει να μην γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Η αρχική αντίδραση στο δικό μας το έργο και άλλων ήταν να ε, πείσουν ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι, να μας θεωρήσουν αναξιόπιστους. Όμως δεν γινόταν. Προσπάθησαν να μας υπονομεύσουν με διάφορους τρόπους, λέγοντας ότι το NDC είναι καλύτερο γιατί είναι ε, ίδιο για όλους, για παράδειγμα. Ίσως και συνείδητα να υπήρχε επιθυμία να μην πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Να μην χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν. Εγώ δεν ξέρω να έχει υπάρξει κάποια συλλογική δράση, κάτι επίτηδες, αλλά ε, συλλογικά ότι ασυνείδητα άφησαν ε, το πρόβλημα να βρίσκεται χωρίς να το αντιμετωπίσουν, ναι καλύτερα να ασχοληθούμε με άλλα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δηλαδή ότι έτσι αντέδρασαν. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση κυρία Μόλτεν. Εγώ είμαι κάπως κάπως βλέπω να είστε σκεπτικιστή σε σχέση με την πρόοδο των εκπομπών για τα οξύδια ζώτου γιατί όμως λέτε ότι υπήρξε μια βελτίωση μεταξύ των Euro 5 και Euro 6, μια βελτίωση στις εκπομπέ NOx. η οποία έχει να κάνει με την ε, επικείμενη εφαρμογή δοκιμασιών σε πραγματικές συνθήκες, πιστεύετε ότι αυτή είναι η σύνδεση, αυτός είναι ο λόγος που υπήρξε η βελτίωση. Υπήρξε βελτίωση τις ε, ε, εκπομπές σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μεταξύ γύρω 5 και γύρω 6 περίπου με, με τα ε, περίπου μείωση στο μισό των εκπομπών σε πραγματικές ε, συνθήκες. Αυτό το οποίο δεν υπήρξε ήταν βελτίωση στον παράγοντα συμμόρφωση. Τέσσερις φορές ήταν για, τον, για το Euro 5 και τέσσερις φορές για το Euro 6, οπότε δεν υπάρχει βελτίωση. Σε πραγματικούς όρους έχουν μειωθεί οι εκπομπές. Και αυτό οφείλεται βέβαια και στους κανονισμούς του Euro 6, αλλά επίσης και τον κίνδυνο, την απειλή ότι θα γίνουν πιο σκληρές οι δοκιμές λόγω των δοκιμών σε δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες. Βέβαια, έχουμε κάποια οχήματα τα οποία μπαίνουν πρώτα στην κατηγορία Euro 6 είναι από τις κατασκευαστές που έχουν τις καλύτερες τεχνολογίες για τη μείωση των οξυδίων του αζότου. Μπορεί ο παράγων αυτός να ξαναανεβεί. Γιατί ακόμα και αυτοί που δεν έχουν την καλύτερη τεχνολογία πρέπει να φέρουν τέτοια αυτοκίνητα στην αγορά που να ανήκουν στην κατηγορία Euro 6. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε τόσο πολλές φορές πάνω από το όριο στα Euro 6 όσο ήμασταν στο Euro 5. Φυσικά το, οι πραγματικές ε, εκπομπές έχουν μειωθεί. Ευχαριστώ κύριε Μόρδεν Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους υπήρξαν πληροφορίες στον τύπο που είπαν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, μιμηθεί την ευρωπαϊκή μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της κατανάλωσης των καυσίμων. Αυτό ισχύει και για τις εκπομπές. Και γιατί υπήρξε αυτή η δήλωση, δεν το κατάλαβα αυτό. Έκαναν κάτι τέτοιο δεν. Δεν ενθυμούμαι εγώ γενικότερα. Πάντως οι Αμερικανοί κάνουν τις δικές τους διαδικασίες και τις κάνουν σχετικά γρηγορότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν παράδειγμα, όταν περνούν από το FTP 75 στο νέο κύκλο δοκιμών με πέντε ε, διαδοχικούς κύκλους, το έκαναν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να καλύψουν ακριβώς τις διαφορές που είχαν στις ε, υποδήλωση εκπομπές και στις πραγματικές εκπομπές. Χρησιμοποίησαν λοιπόν τους συμπληρωματικούς κύκλους δοκιμών για να κλείσουν το κενό. Και σήμερα δεν υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπει στις επικολούμενες ετικέτες ο Αμερικανός οδηγός και σε σχέση με αυτά τα οποία δημοσιεύονται μετά από τους ελέγχους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν προχώρησαν πιο γρήγορα και πιο επιθετικά και για τις εκπομπές και για την κατανάλωση. Αντίθετα λοιπόν, εδώ λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρωτοπόρος σε σχέση με την κατανάλωση και σε σχέση και με τις πραγματικές εκπομπές είμαστε στα υψηλότερα, στα καλύτερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Πώς συνδυάζεται αυτό με αυτό το οποίο είπατε εσείς. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν, αυτές αν αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα του αυτοκίνητο, της αυτοκίνητοβιομηχανίας. Και η νέα κατάσταση η οποία δημιουργείται σε σχέση με τις ε, νέες μορφές ελέγχου θα βελτιώσει τις πληροφορίες οι οποίες δίδονται στους καταναλωτές που εσείς είπατε ότι είναι ελληματικοί. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε φυσικά ότι οι καταναλωτές δεν είναι και όλοι μηχανολόγοι. Ε, βέβαια, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εισαγωγή των PEN στο σύστημα ελέγχου τύπου πρωτοπορεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Το αμερικανικό σύστημα δίδει την έγκριση τύπου στο εργαστήριο, αλλά χρησιμοποιούν τα PEMS, τους κινητούς ελέγχους, ε, για ε, την επαλήθευση των επιδόσεων. Ε, το κάνουν λοιπόν σε επίπεδο εργαστηρίου, αλλά είναι πιο απαιτητικοί και επιθετικοί. Εμείς σε επίπεδο έρευνας λοιπόν καθοδηγούμε μεν, αλλά όχι προς τη σωστή κατεύθυνση πάντα. Δεύτερη ερώτηση, η ανταγωνιστικότητα <clears throat> της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Κατά κάποιο τρόπο, και μπορεί αυτό να ισχύει, ότι στόχος ακριβώς των ρυθμίσεων είναι να δημιουργούν ένα επίπεδο ισοτιμίας. Αυτό που δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα είναι όταν ένα επίπεδο ισοτιμίας δεν ισχύει πλέον. Έχουμε να κάνουμε με μια ονομαστική ισοτιμία σήμερα. Κάποιοι κατασκευαστές παίζουν με τις ρυθμίσεις περισσότερο από άλλους και αποκτούν πλέον εκτήματα ανταγωνιστικότητας ως μειόφυλαν. Συνεπώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ε, σε επίπεδο εξαγωγών δεν τίθεται πρόβλημα, νομίζω, γιατί μπορούν ε, τα προϊόντα να διαφοροποιούνται μετά από την ε, παράδοση και πώληση ή μπορεί και να μην έχουν. Λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό το να υπάρξει απώλεια ανταγωνιστικότητας. Το θέμα είναι να υπάρχει δικαιοσύνη σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας στην Ένωση. Ε, καλύτερη ενημέρωση στους καταναλωτές. Δυνητικά ναι, θα πρέπει να γνωρίζουν τι δημοσιεύεται, με ποιο τρόπο, με ποιο χρονισμό και με ποιο επίπεδο λεπτομέρειας. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε και το δίκτυ Aqua, ο οποίος σε καθημερινή βάση δείχνει το τι συμβαίνει στους καταναλωτές είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά. Εμείς θέλουμε να συμβουλεύουμε με απλό τρόπο τους καταναλωτές. Και νομίζω ότι τα νέα στοιχεία, τα επίσημα θα βοηθήσουν και αυτά. Αλλά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και νομίζω ότι κατά 99,9% οι καταναλωτές δεν θα είναι σε θέση να τα ερμηνεύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε που είσαστε ενώπιον μας να ανταλλάξουμε απόψεις. Λέτε στην ιστοσελίδα σας ότι η τεχνολογία αυτή PEMS είναι εδρεωμένη και χρησιμοποιείται ήδη από δημόσιες αρχές. Ποιος το κάνει αυτό όμως. Και επίσης είπατε ότι πληροφορήθηκαν οι κυβερνήσεις για τα θέματα αποκλήσεων μεταξύ των πραγματικών εκπομπών και των εκπομπών στη, στο εργαστήριο, αλλά δεν έχουν αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Οι κύριοι χρήστες των ΠΕΜΣ e ήταν οι Αμερικανοί και πράγματι εισήχθη στις Ηνωμένε Πολιτείες μετά από τη χειραγώγηση τέλο πάντων από το θέμα ακριβώς των παρακαπτικών εξοπλισμών στα τέλη της δεκαετίας του 90. Που ήταν λίγο πολύ ότι έκανε και Volkswagen. Τα PEMS λοιπόν δημιουργήθηκαν ακριβώς για να ελέγχουν τα φορτηγά σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Οπότε η τεχνολογία ε, υπήρξε κατά κάποιο τρόπο ήδη εδώ και αρκετό καιρό μέχρι από πριν από πέντε χρόνια ήταν ε, απλώ και μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Καλιφόρνια που χρησιμοποιούνται εκεί είχαν το περισσότερο εξοπλισμό για αυτά τα PEMS και τα χρησιμοποιούσαν εκεί. Και μάλιστα κοιτάζαν να δούνε και σε τι βαθμό λειτουργούσαν καλά. Ε, δεν νομίζω εκτός από τις ΗΠΑ ε, χρησιμοποιόντουσαν μόνο όταν αρχίσαμε εμεί στην Αγγλία να τα χρησιμοποιούμε. Βέβαια, ίσω η αυτοκινητοβιομηχανία ε, πίσω από κλειστέ πόρτε. Αλλά πόσο ξέρω, μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά μα είπαν οι εμπειρογνώμονε ότι υπάρχει μια βεβαιότητα 30% στι μετρήσει. Αυτό ισχύει για την τεχνολογία πέμψη, όχι. Εγώ έχω μια κάπως διαφορετική άποψη, βασιζόμενος αποκλειστικά στα δικά μας τα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι αν κάνεις ε, μία δοκιμή ενόξου οξυδίων σε πραγματικές συνθήκες, συν πλήν 25% θα έχεις αποτέλεσμα αξιοπιστίας. Αν κάνεις μια αντίστοιχη δοκιμή σε ένα φορτηγό, σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς όμως ε, να εξαρτάται από την κίνηση, τότε θα πάρει σαν αποτέλεσμα ένα συν πλήν 10% αξιοπιστία. Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική βέβαια από τις προφορίες που έχουμε το JRC που μιλάει για 30% μεταβλητότητα. Εξαρτάται βέβαια από την ανάλυση που γίνεται. Αν σταθμίσετε τα αποτελέσματα, το έχετε και κάποια διόρθωση που μπορεί να μειώσει το βαθμό μεταβολής σε σημαντικό βαθμό. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει κανείς για να βελτιώσει το μεταβλητό των δοκιμών. Μπορείτε να κάνετε καλά δοκιμές πέμψη και μπορείτε να τις κάνετε και στραβά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να διασφαλίζουμε ότι γίνονται καλά οι δοκιμέ αυτές τις πέμψεις. Και αν γίνονται καλά, τότε το μεταβλητό των δοκιμών αυτών είναι κάτω από 10%. Θέλετε να αναπτύξετε λοιπόν και μεθόδου, προτάσει για το πώ να χρησιμοποιείτε τη τεχνολογία πέμψη. Ένα πρακτικό θέμα τώρα για τι δοκιμασίε που κάνετε. Έχετε 500 αυτοκίνητα που δοκιμάζετε κάθε χρόνο. Πώς τα παίρνετε αυτά τα αυτοκίνητα, τα αγοράζετε, τα νοικιάζετε, σας τα δίνουν κατασκευαστές. Πώς τα επιλέγετε αυτά τα αυτοκίνητα που δοκιμάζετε. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μην φτάσουν στα χέρια μας οχήματα τα οποία να είναι πειραγμένα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε έχουμε διαφορετικές πηγές. από μέσα ενημέρωσης δημοσιογράφων δηλαδή, αλλά και άλλα μεταχειρισμένα. Οι μερικές φορές μάλιστα αγοράζουμε και οχήματα. Έχουμε δηλαδή ποικιλία πηγών που προμηθευόμαστε. Μερικά τα αγοράζουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά ποτέ δεν ανακοινώνουμε αποτελέσματα, δεν έχουμε δοκιμάσει και ένα άλλο αντίστοιχο όχημα εντελώς ανεξάρτητα. Ποτέ δεν έχει πέσει πάντω στα χέρια μας κανένα πειραγμένο. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο εύρος πηγών από τις οποίες προμηθευόμαστε τα οχήματα ακριβώ για να είναι ανεξάρτητα τα αποτελέσματά μας. Κύριε Ριβό, ευχαριστώ. Μια που απαντήσατε στις άλλες ερωτήσεις, θέλω να ρωτήσω κάποιες διευκρινήσεις, όχι για τα πέμψε, για τα άλλα είδη δοκιμών που γίνονται. Τι γνωρίζετε για αυτά τα άλλα τεστ, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα με λέιζερ ή τηλεμετρία. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για τέτοιου είδους δοκιμές. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, λέτε ότι υπάρχει μια εναλλακτική εξοπλισμού PEMS που βασίζεται στην τεχνολογία laser, τα FTR. Και το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί ταυτόχρονα να μετρήσει πολύ περισσότερες ρηπογόνες ουσίες. Είναι πολύ υποσχόμενος ο εξοπλισμός αυτός και πολλές δυσκολίες έχουν ήδη ξεπεραστεί. Όπως για παράδειγμα το μέγεθος, η κατανάλωση, το βάρος. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες μονάδες από μια ιαπωνική εταιρεία που όμως ζυγίζουν το διπλό από τον εξοπλισμό PEMS που διαθέτουμε τώρα. Δεν έχει μέσα το flow tube που είναι κάτι πολύ βασικό για την ρύθμιση των δοκιμών. Η τεχνολογία είναι πολύ υποσχόμενη αλλά δεν είναι ακόμα υπαρκτή για μας προς χρήση. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε την ενέργεια του οχήματος γιατί τότε θα λιώνεται ε, ακριβώς το τεστ. Οπότε δεν θέλουμε έναν βαρύ εξοπλισμό, γιατί τότε θα πρέπει να το λάβουμε και αυτόν υπόψη μας. Δεν επιτρέπεται όμως. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η τεχνολογία χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να είναι χρήσιμη. Πάντως είναι ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά θετικά. Όπως σας είπατε, ταυτόχρονα ε, μετράει τις λιπογόνες ουσίες πολλών διαφορετικών ε, ρήπων. Στην ερώτηση 4 απαντήσατε για κύκλους δοκιμών στο εργαστήριο όπως είναι το θερμικό παράθυρο. Τι άλλου είδους τέτοιες δοκιμές γνωρίζετε, πού βασίζονται και πού κινδυνεύει να υπάρξει κύκλωμα. Το πρόγραμμά μας δεν το έχουμε ετοιμάσει για να αντιμετωπίσουμε τους παρακαμπτικούς αυτούς εξοπλισμούς. Όχι, δεν έγινε για αυτό το σκοπό. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή η Volkswagen τι έκανε, κάτι ασυνήθιστο και περιτά περίπλοκο. Το να φουσκώνει τα λάστιχα έχει μεγάλο όφελος. Η άλλη στρατηγική που πολύ εύκολη είναι και μπορεί να γίνει με τεχνολογία όχι ιδιαίτερα εχμής. Υπάρχουν πολύ εύκολοι τρόποι για να βελτιώσει κανείς τα αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται αλγόριθμους ή άλλα περίπλοκα λογισμικά. Το θέμα αυτό των θερμικών παραθύρων που λέτε είναι ένα σύστημα που χρειάζεται περίπλοκους αλγόριθμους, αλλά είναι ένα σχετικά απλό σύστημα, το συγκρίνουμε με αυτό που χρησιμοποιεί η Volkswagen. Και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα θερμικά παράθυρα και ότι η αυτοκινητοβιομηχανία τα χρησιμοποιεί συχνά. Εμείς έχουμε κάνει δοκιμές σε διάφορες θερμοκρασίες, σε πολλά οχήματα, από 5 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλύσαμε τα στοιχεία πάνω και κάτω από αυτά τα όρια της θερμοκρασίας για να δούμε ε, οι μέση όροι της αυτοκινητοβιομηχανίας τι διαφορές έχουν. Λίγες περιπτώσεις ξεχωρίζουν και αυτό δείχνει ότι μάλλον χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική, την στρατηγική στην οποία αναφερθήκατε. Μια ακόμα ερώτηση. Πιστεύετε ότι τεχνικά είναι εφικτό να βασιστούμε στα στοιχεία που έχουμε από τα ΟΜΠΕΝΤΕ για να εκτιμήσουμε χοντρικά τις εκπομπές και μετά να τις συγκρίνουμε με τις πραγματικές ώστε έτσι να καταλήξουμε σε δείχτες ε, και να καταλάβουμε κατά πόσο οι δοκιμές στη μία και στην άλλη περίπτωση ισχύουν ή όχι. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά έχουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν μπορούν με τίποτα να υποκαταστήσουν ανεξάρτητους ελέγχους ή πιστοποίησεις. Δεν ξέρετε πόσο έγκυρα είναι τα στοιχεία OBD και για να το μάθετε αυτό, τότε χρειάζεστε μια ανεξάρτητη έρευνα που απαιτεί πάλι έναν ε, σύνθετο εξοπλισμό. Άρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Δεν βοηθάει καθόλου αυτό on-board diagnostics. Μιλάμε λοιπόν για γενικές τάσεις. Κατά μέσο όρο, κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε ή μειώνουμε τα οξύδια του αζότου, ναι, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ελέγχους. Ο κύριος Δεσμάκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ολλανδικά, επιτρέψτε μου. Η Mission Analytics είναι μια οργάνωση λοιπόν η οποία κάνει ίδια δοκιμές και έχει επιφέρει κριτική και στην αυτοκινητοβιομηχανία για τους τρόπους και τη μεθοδολογία των δοκιμών που διαφέρουν τόσο πολύ ώστε τα συμπεράσματα δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα. Άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Τι λέτε εσείς για την κριτική αυτή. Μιλάτε το ότι ακριβώς είναι πολύ διαφορετικά τα αποτελέσματα, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα έχω να προσάψω στη μεθοδολογία αυτή. Ο... Η αυτοκινητοβιομηχανία έρχεται λοιπόν με τα δικά της στοιχεία βάσει κάποιων προδιαγραφών. Κατά τη γνώμη μου μπαίνει πολύ μεγάλο βάρος στο σκέλος τυποποίησης ενώ θα έπρεπε η τυποποίηση να είναι από την αρχή. Γι' αυτό οι δοκιμές που κάνουμε εμείς κάθε φορά ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με το δικές μας τις προδιαγραφές και τη δικιά μας τη στρατηγική. Δεν υπάρχουν εκεί μεταβλητές και δεν βασιζόμαστε σε στατιστικές. Γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε μεγάλες διαφορές κι εμείς. Υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα στο σύστημα που μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε κεντρικά να το κάνουμε και ελεγχόμενα, γιατί ναι, υπάρχει βέβαια κάποια, κάποιο στοιχείο μεταβλητού, αλλά θέλουμε αυτό να το ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Από την αρχή, από την μορφή, από τις συνθήκες. Έτσι ώστε τα εργαλεία τυποποίησης να επηρεάζουν όσο γίνεται λιγότερο το αποτέλεσμα. Είναι μια αδυναμία στο... στα δεδομένα αυτά ότι Στην απάντησή σας στην ερώτηση 3 λέτε ότι τεχνικά είναι δυνατόν τα οχήματα diesel να προσαρμοστούν, να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέτε ότι το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία επιλέγει τα οξύδια του αζότου μπορεί να καταλήγει σε ένα πρόβλημα τυποποίησης και ότι η ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκεί. Σε άλλες ε, ερωτήσεις απαντάτε με τον ε, ε, δείκτη συμμόρφωσης και στην απάντησή σας στην ερώτηση 9 λέτε ότι επιλέγετε το 2,1 γιατί μπορεί να επιτευχθεί με ένα απλό λογισμικό του, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εσείς τι παραπάνω μπορείτε να μας πείτε ώστε να μην υπάρχει διαφορά στην εφαρμογή. The key thing to... Το ουσιαστικό συστηματικό στοιχείο του, των ε, πραγματικών δοκιμασιών είναι και το σύστημα εποπτείας για τις ε, δοκιμές αυτές. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρο πέφτει στην έγκριση τύπου. Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Το RDE μα δίνει δυνατότητα να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα έγκρισης τύπου και τα ασφάλματά του μπορούν να αντισταθμιστούν από, μια αυστηρή, ε, από ένα αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθηση ενό αυτοκινήτου όταν λειτουργεί. Γιατί φυσιολογικό είναι να θέλουν οι κατασκευαστές να μειώσουν στο δυνατό λιγότερο την, ε, την, ε, τις εκπομπές που μετρούνται για τα οξύδια, γιατί όλα αυτά, για, να μειώσουν τις εκπομπές, αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Μειώνει την ε, ισχύ του αυτοκινήτου, αυξάνει το κόστος κτλ. Κανείς δεν θέλει να τα κάνει αυτά. Δεν υπάρχουν εύκολοι, είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς τρόπους να παρακάμψει το σύστημα Έγκριση τύπου, ενώ αν υπάρχει μια δυνατότητα να παίρνει κάνει στοιχεία αυτοκίνητα από το δρόμο και να τα εγκρίνει με τον τρόπο αυτό, ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει, ακόμα και αν κάνει κανεί κόλπα εκεί πέρα, όταν ελέγχει στην τύχη αυτοκίνητα στον δρόμο, ξέρει ότι εκεί πέρα θα τον πιάσουν. Η κυρία Χίρινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να προτιμάει την εφαρμογή του LNT αντί του SRC, SR, Ευρώ 6. Το Ευρώ 5 και Ευρώ 6 θα μπορούσαμε να τα προσαρμόσουμε μόνο με το LNT και μπορεί να υπάρξει συνδυασμός του LNT και του EGR αντί να αντικατασταθεί εντελώς το LNT από το EGR. Γίνεται. Τα πρότυπα Euro 6 μπορούν να επιτευχθούν μαζί με τη χρήση του συστήματος επανακυκλοφορίας των καυσαερίων και με τα λεγόμενα Lean NOx traps, με τις παγίδες οξυδίων. Εμείς ε, δώσαμε αλφα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ε, τέσσερα αυτοκίνητα τα οποία τηρούσαν τις προδιαγραφές και τέσσερα από αυτά είχαν τα συστήματα LNT. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη το LNT γιατί το πρόβλημα με το LNT είναι υπάρχει κάποιο όριο για το πόσο πόσα οξύδια ζώτου μπορεί να συγκρατήσει. Αν είναι πιο αυστηροί οι κανόνες στο μέλλον, εγώ φοβάμαι ότι οι κατασκευαστές δεν θέλουν να έχουν επενδύσει στην τεχνολογία LNT και η τεχνολογία αυτή φτάνει σε κάποιο όριο και πρέπει να πάνε σε κάποια άλλη τεχνολογία όπως η τεχνολογία SCR. Ίσως είναι καλύτερα να πάμε τώρα στο SCR γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα ε, να μειωθεί σημαντικά η εκπομπή οξυδίων του, του αζότου. Ίσως είναι η, το όριο του LNT ότι μπορεί τώρα να λύσει το πρόβλημα, αλλά ενδεχομένω θα προτιμήσουν οι κατασκευαστέ να πάνε στην επιλεκτική μείωση, καταλητική μείωση, γιατί το SCR, γιατί στο μέλλον έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη. Ευχαριστώ. Έχω άλλη μια ερώτηση. Στην απάντησή σας στην ερώτηση 10 λέτε ότι από τα 8 οχήματα, από τα 8, από ναι, που, που είχαν πρόβλημα με τα πρότυπα Euro 6, τα 7 ήταν της Volkswagen. Πώς μπόρεσαν να τηρήσουν τις προδιαγραφές, γιατί τα 7 στο 8 μπόρεσαν να τα τηρήσουν και γιατί το 1 δεν τα μπόρεσε να πετύχει τις προδιαγραφές, να θεωρηθεί ότι πέτυχε στη δοκιμή. το μέγεθος και η μορφή του κάθε συστήματος παίζει ρόλο. Τέσσερα συστήματα είναι αυτά που μερικές φορές ξεπερνάνε 20 φορές τα όρια. Και με το LNT το ίδιο ισχύει. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν φτιαχτεί τα συστήματα αυτά. Για το LNT ποιες είναι οι στρατηγικές και για το ECR ποιο είναι το ποσοστό έγχυσης. Αν τα χρησιμοποιήσετε διαφορετικά, έχετε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Η έγχυση αυτή είναι το σημαντικό. Για το SCR υπάρχει μια εύκολη λύση. να αρχίσεις περισσότερο, δουλειά. μερικέ φορές μπορεί να είναι αυτή η λύση. Υπάρχει όφελος και ζημία κάθε φορά. Γι' αυτό και δεν το κάνεις παρά μόνο αν πρέπει να το κάνεις. Αλλά σίγουρα για το SCR e είναι πολύ εύκολο να το ανοίξει να το κλείσεις το σύστημα όπω θέλει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βίλξ. Ο κύριος Έκχαουτ είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντεν που μας εξηγήσατε τις διάφορες τεχνολογίες και εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο περισσότερο για τις τεχνολογίες αυτές ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι τεχνικά εφικτό και πού βρίσκονται τα όρια. Εσείς κάνετε μετρήσεις και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εγώ κοιτάζω μονάχα τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα δίζελ. Ξέρουμε ότι στις Ηνωμένες τα πρότυπα είναι διπλάσια σε αυστηρότητα από την ε, Ευρώπη, δηλαδή το επίπεδο είναι το μισό της Ευρώπης και της Καλιφόρνια είναι πολύ χαμηλό, είναι ακόμα χαμηλότερο. Λέτε ότι μπορεί ακόμα και με την τωρινή τεχνολογία, συνδυάζοντας το LNT και το SCR, e να πετύχουμε ακόμα και τα πρότυπα της Καλιφόρνιας να ε, τηρήσουμε. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα αμερικανικά όρια είναι 31 μιλογκράμμ για χιλιόμετρο σε σχέση με τα δικά μας 80, κάτω από το μισό. Στα πετρελαιοκίνητα που πολλούνται εδώ και χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείε καλύπτουν το όριο αυτό μόνο με το σύστημα SCR. Η BMW συνδυάζει το LNT και το SCR για να αντιμετωπίσει εν μέρη την αδυναμία του SCR που είναι οι υψηλές εκπομπές NOx όταν είναι κρύος ο κινητήρας. Στην διαδικασία θέρμανσης του κινητήρα δηλαδή δεν λειτουργεί το SCR. Ερώ το τι λειτουργεί καλά και σε αυτή τη φάση. Οπότε έχουν και τους δύο μηχανισμούς για να καλύψουν όλους τους κύκλους λειτουργίας του κινητήρα. Έρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Αυτό το οποίο δεν θέλει κανείς σαν κατασκευαστής είναι να τον πιάσουν στο μέλλον ότι δεν σέβεται τα όρια. Βάζοντας και τους δύο μηχανισμούς τότε καλύπτει στο σύνολο του προβλήματος. Μπορούν να το κάνουν βέβαια και μόνο με το SCR, αλλά είναι λίγο πιο επικίνδυνο, λίγο πιο αβέβαιο. καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό κάνει το αυτοκίνητο πιο ακριβό. Γι' αυτό τα γερμανικά ντίζελ στις Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούνται πολυτελείας και είναι πιο ακριβά κατά εκατοντάδες δολάρια. Βέβαια αυτό είναι ένα χαμηλό τίμημα γιατί δεν θα ήθελε κανείς να συλληφθεί μη σεβόμενο στις ρυθμίσεις της Καλιφόρνια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την ίδια αγορά με τη ΣΥΠΑ, οπότε η ανταγωνιστικότητα φύγει όλους τους βιομηχάνους, τους αυτοκινητοβιομηχάνους. Για να το πω λίγο πιο απλά, σε επίπεδο τεχνικό υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες που μπορούν να καταστήσουν τα ευρωπαϊκά στάνταρτς απόλυτα εφικτά. Φυσικά, απολύτως οι ρυθμίσεις για τον όξο στην ΕΠΑ καλύπτονται από τους Γερμανούς καταναλωτές εδώ και χρόνια με τις ίδιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Γενικά το λέω αυτό αλλά με έγχυση ουρία σε υψηλότερη δοσολογία από ό,τι το κάνουν στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη προσπαθούν αυτό να το ρυθμίζουν κάθε φορά που κάνει σέρβι το αυτοκίνητο, αλλά στην ουσία όσο χρησιμοποιείς ουρία τόσο α, μειώνεις τον όξο. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες διαθέσιμες, οι οποίες δεν είναι εφαρμογή στα επιβατηγά όπου μπορεί κανείς να πέσει ακόμα πιο πολύ. Υπάρχουν συστήματα σαν παράδειγμα έγχυσης καθαρής αμμονίας η οποία μπορεί να αποθηκεύεται ε, με στερεή μορφή μέσα σε ε, φορείς μεταλλικούς και αυτό να αναμειγνύεται με τη ροή εξάτμισης και να κόψεις έτσι το 98% το οξύδιο του αζότου. Αλλά νομίζω ότι η χρήση της ουρίας νομίζω ότι ε, είναι ένας δρόμος και επελέγει για ιστορικούς και εμπορικούς λόγους από τη χρήση της αμμονίας. Υπάρχει τεχνολογία, χρησιμοποιείται σε λεωφορεία κτλ. Λοιπόν, χωρίς να εφεύρουμε οτιδήποτε νέο, μπορούμε να κόψουμε όσο περισσότερο νόξ θέλουμε. Το θέμα είναι διακανονιστικό πόσο θέλουμε να μειώσουμε τον όξ και με τι τίμημα. Να δούμε ποιο είναι το κόστος λειτουργίας και για τον καταναλωτή. Η πολιτική επιλογή πρέπει να γίνει, η δυνατότητα υπάρχει. Τότε γιατί εμείς σαν υπεύθυνοι έχουμε αποφασίσει το 2,1 παράγοντα συμμόρφωσης, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Η άποψή μου γι' αυτό είναι η εξής. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές επιδόσεων ανάμεσα στους, κατασκευαστές. Πολλοί από αυτούς μπορεί να πετύχουν εύκολα το 1,5 ή Volkswagen ή BMW ε, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν στον ίδιο χρόνο. Και γι' αυτό λοιπόν υποπτεύομαι ότι η λύση που δόθηκε είναι γιατί δεν ήξεραν πόσο σίγουρη ήταν η τεχνολογία τους. Ξέρατε όμως ότι τα επίπεδα είχαν ήδη από το 2007. Το θέμα είναι πώς θα προσπαθούσαν να τα επιδιώξουν και με ποιο βαθμό τα δεδομένα θα μπορούσαν, κάποιοι από αυτούς πίστευαν, να υπονομεύσουν, να αποδυναμώσουν, να βρουν παραθυράκια, αλλά αυτό τώρα είναι μια υποψία, δεν έχω τεκμηρίωση γι' αυτό. Το σκέφτηκαν όμως γιατί είχαν σκεφτεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν ε, και δεν θέλησαν να επενδύσουν επίσης. Και ξαφνικά συμβαίνει το Dieselgate και δίδεται μια πολιτική όθηση και τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι βλέπω εγώ την κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ξεκινάμε τον δεύτερο βέβαια. Ανά τρεις ε, ε, ερωτήσεις. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. έτσι ώστε να υπάρξει χώρος για να δοθούν απαντήσεις. Ο κύριος Μπελέτ έχει το λόγο. Δίπλα σας είμαι κύριε Μόλτεν. Θα ήθελα να επανέλθω στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα όρια των εκπομπών. Είναι μιλιγράμμα ένα χιλιόμετρο, αλλά βάσει της έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών, λέει στην έκθεσή του το κέντρο, στην έκθεση του 2011 ότι αυτή η μέθοδος έκφρασης των ορίων αυτών είναι προβληματική γιατί δεν υπάρχει αναφορά στις ε, παραμέτρους του κινητήρα <clears throat> και δεν λαμβάνει υπόψη αυτή η έκφραση την ε, μεταβλητότητα επί τη βάση των διαφορετικών συνδικών στον δρόμο μπορείτε να πείτε αν εσείς συμφωνείτε με αυτές τις ε, διατυπώσεις και πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να εκφράσουμε την, ε, τις εκπομπές. Λοιπόν, η σύντομη απάντηση ίσως είναι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. <clears throat> Τι γίνεται με τα αυτοκίνητα, με τα μεγάλα φορτηγά, είναι ε, μιλιγκράμμ ανά κιλοβατόρα, δηλαδή η μονάδα έργου που κάνει το μηχάνημα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπορείς κάτι να μετρήσει κάτι τέτοιο με τα οχήματα αυτά. Ας πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, αλλά όταν έχουμε όλα τα είδη <clears throat> επιβατικών αυτοκίνητων που θέλουμε να δοκιμάσουμε είναι πολύ πιο δύσκολο. Και δεν θέλετε να βασίζετε μονάχα στο ε, μήνυμα που σας δίνει ο υπολογιστής του αυτοκίνητου που μπορεί να, έχει, να το έχει μαγειρέψει ο κατασκευαστής. Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρούμε ένα μέτρο του έργου που καταναλώνει το αυτοκίνητο που είναι ανεξάρτητο από το ίδιο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό μπορεί κανείς να μετρήσει τις ε, εκπομπές ανεξάρτητα από το όχημα και την απόσταση που διανύει με GPS, επομένως δεν μπορεί ο κατασκευαστής να σας γελάσει. Βέβαια, είναι πραγματικότητα ότι ο κινητήρας χρησιμοποιεί πιο πολύ, καταναλώνει πιο πολύ έργο όταν ξεκινάει και σταματάει κάθε τόσο κανείς. Αλλά το θέμα είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ιαπωνία προσπαθούν να βρουν ένα νέο επιστημονικό τρόπο να λύσουν αυτό το πρόβλημα ακριβώς για να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους οι οποίες διακυμαίνονται και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα μέθησης. Δεν ξέρω αυτά που έχουν γίνει για την αλλαγή του τρόπου μέθησης. Μα το καλύτερο είναι να έχετε διαφορετικούς ε, τομείς μέτρησης ε, στην πόλη, στο δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό δεν είναι πιο κομψή λύση, αλλά είναι πρακτική λύση. Δεν έχω, δεν έχω βρει να υπάρχει κάποια άλλη ε, βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Σούλτσε. Ο κύριος Σέρτουκ είναι πρώτα. Και μετά ο κύριος Σούλτσε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Μόλτε, να επανέλθω αυτά που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι ήσασταν σε επαφή με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί αναφερθήκατε στις αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν <clears throat> μεταξύ ε, εργαστηρίου και δρόμου. Μιλήσατε για αυτά με τις αρχές σας. Εμείς έχουμε δημοσιεύσει πληροφορίες δημόσια, έχουμε μιλήσει σε συναντήσεις, σε συνδιασκέψεις. Εμείς έχουμε μιλήσει με οποιονδήποτε θέλει να μας ακούσει από το 2012. Και το τελευταίο χρόνο υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση του Ρωμαίου Βασιλείου και από άλλες κυβερνήσεις αλλά υπήρξε πρόβλημα αξιοπιστίας όταν κατάλαβαν όλοι ότι αυτό που λέγαμε ότι είναι τέσσερις φορές πάνω από τα όρια ε, ότι αυτό βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Εμεί προσπαθούσαμε να μιλήσουμε σε όλου, να πούμε να εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα, να έχουμε μια νέα μεθοδολογία. Ακούστε σε αυτό που, αυτό που σα λέμε. Κάποιοι μα άκουσαν, κάποιοι όχι. Λέτε ότι σα άκουσαν όλοι. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιε ήταν οι αντιδράσει από τη στιγμή και πέρα που άρχισαν να σας ε, ακούνε. αυτό εξαρτάται από το συνομιλητή μας. Από την πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανίας η απάντηση ήταν «Ε, εντάξει, αλλά χρειαζόμαστε ένα τεστ το οποίο θα είναι σωστό για όλους, ε, γιατί μόνο στο εργαστήριο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, το PEMS δεν είναι, ακρι, δεν είναι πολύ ακριβές. Μόνο το Dieselgate άλλαξε την ιστορία, το, το αφήγημά τους. Αυτή ήταν η απάντηση της βιομηχανίας. Και οι κυβερνητικοί φορείς στους οποίους μιλήσαμε, οι περισσότεροι, σε μεγάλο βαθμό ακολουθούν αυτά τα οποία θέλουν οι βιομηχανοί. Ένα τελευταίο ερώτημα προτού τελειώσει ο χρόνος. Στην απάντηση για το ερώτημα 9 μιλήσατε για ένα de facto παράγοντα συμμόρφωσης 0,4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς έχετε φτάσει σε αυτή την εκτίμηση και πού είναι οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σε σχέση με τον παράγοντα συμμόρφωσης. Ε, το θέμα είναι και σε επίπεδο διακανονιστικό, δηλαδή εδώ έχουμε 80 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο στην Ευρώπη, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι 35. Συνεπώς λοιπόν, 31 μάλλον, βλέπετε ότι έχουμε μια, έναν λόγο διαφορά σημαντικό. Και δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα βέβαια, γιατί οι δοκιμέ γίνονται με διαφορετικό τρόπο, αλλά παρόλα αυτά το ανώτατο όριο είναι σε μάσα δηλαδή, υπερδιπλάσιο του Αμερικανικού και αυτό κάνει εντύπωση. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Έχω δύο ουσιαστικά ερωτήματα. Ένα βασίζεται σε μία απάντηση που δώσατε πριν από λίγα λεπτά είπατε ότι η Volkswagen και η BMW θα μπορούσαν χωρίς κανένα πρόβλημα να πετύχουν το 1,5 ως παράγοντα συμμόρφωσης, ενώ άλλοι κατασκευαστές όχι. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, το λέτε αυτό επειδή ξέρετε αυτούς τους δύο κατασκευαστές. Μπορείτε να πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Εγώ μπορώ να σας δώσω ονόματα, λέει ο κ. Μόλτον. Έχουμε κάνει μελέτες με αντίστοιχους φορείς στην... Proved that the Volkswagen Golf um, was the cleanest of the lot by, by some margin. Uh, the dirtiest vehicle... Χωρίς μικρόφωνο Εκεί που ήθελα να πω το όνομα, κόπηκε το μικρόφωνο. Το Fiat 506 ήταν το πιο βρώμικο από τα αυτοκίνητα που δοκιμάσαμε. Περίπου 10 φορές το όριο. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα δοκιμάστηκαν στην ίδια διαδρομή, την ίδια εβδομάδα από τους ίδιους οδηγούς. Το Volkswagen ήταν μια μισή φορά περίπου παράγοντα συμμόρφωση και το Fiat 10. Όλα αυτά ήταν αυτοκίνητα που είχαν εγκριθεί στην κατηγορία Euro 6. Και όχι μόνο το Fiat, υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα που είχαν αρκετά υψηλά, υψηλό παράγοντα συμμόρφωση. Και κάποια οχήματα του ομίλου Volkswagen. Ένα Audi A8 3 λίτρο είχε πολύ ψηλό παράγοντα συμμόρφωση, 20 φορές ήταν ο παράγον συμμόρφωσης. Δεν είναι ότι η Volkswagen είναι τέλειη σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητά σου. Σας δίνει όμως αυτό μια ιδέα του πόσο μεγάλο είναι το φάσμα του παράγοντα συμμόρφωσης. <laughs> Το δεύτερο ερώτημα, και εγώ είμαι μηχανικός, μηχανολόγος. Είπατε ότι είχατε συνεργαστεί με τη Motorsport στη Γερμανία. Πώς εξασφαλίζετε ότι όταν κάνετε αυτές τις ε, μετρήσεις πέμψης δεν μπορούν να γίνονται ε, απάτες. Έχετε ένα μηχάνημα το οποίο μετράει, αλλά πώς ξέρετε εσείς ότι αυτό το μηχάνημα δεν έχει γαργαληθεί, δεν έχει υποστεί χειραγωγήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ελέγχουμε. Οι δύο βασικοί τρόποι είναι οι εξή. Πρώτον, δεν δημοσιεύουμε εμείς τον, με ακρίβεια τον κύκλο δοκιμών και ταυτόχρονα κάνουμε τις δοκιμές στο ίδιο αυτοκίνητο ή περίπου στο ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια στιγμή. Οπότε αν μας έχουν δώσει ένα αυτοκίνητο με επεμβάσεις θα έλεγα, αυτό θα το βλέπαμε στον κύκλο δοκιμών μας στις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί θα είχε διαφορές με το άλλο. Ε, νομίζω ότι είναι ανέφικτο να γίνει κάτι τέτοιο ακόμα και αν κάποιος μας παρακολουθεί από κοντά θα έλεγα για να δει που είμαστε και εμείς κάποια στοιχεία του κύκλου δοκιμών, αν θέλετε, τα αποκρύβουμε έτσι ώστε να μην καθιστούμε διαφανείς τους ελέγχους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι το πρόβλημα των ε, δοκιμών δεν είναι <clears throat> το θέμα τεχνολογίας. Υπάρχουν καλά, καλές δοκιμασίες στο εργαστήριο, υπάρχουν καλές δοκιμασίες στο δρόμο. Αναφερθήκατε τώρα και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγχονται δοκιμασίες που γίνονται σε επιχειρήσεις, στην βιομηχανία. Αλλά είπατε ότι όπως μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ε, παραποιημένα ε, μηχανήματα για το παραπημένες συσκευέ για το εργαστήριο, το ίδιο μπορεί να γίνει να παραπλανήσει κανείς και να τεστ στον δρόμο, έτσι δεν είναι. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να παραποιήσει κανείς μια δοκιμή στον δρόμο με PEMS. Και ο πιο προφανής τρόπος είναι να συγκρίνει κανείς αυτά τα στοιχεία με αυτά που σου δίνει το OBD, το σύστημα του ο υπολογιστής του αυτοκινήτου για τη θερμοκρασία του κινητήρα και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και αυτός είναι ένας τρόπος να λέει στο όχημα ότι αν τώρα με δοκιμάζουν». Και επομένως νομίζω ότι λένε, λέει η νέα οδηγία, δεν πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένο υπολογιστή, ώστε να ξέρει το αυτοκίνητο ότι δοκιμάζεται. Αυτό είναι ένα τρόπο λοιπόν να ξεπεράσουμε ένα κίνητο και κάνουμε και άλλα πράγματα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν μπορεί κανεί να καταλάβει, να ανοιχνεύσει ότι βρισκόμαστε σε δοκιμασία. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχνευτεί μια δοκιμασία PEMS. Και τώρα για το θέμα, ε, είπατε, αυτά που είπατε είναι ενδιαφέροντα πολύ ε, είπατε ότι δεν είναι τεχνικά τα προβλήματα αυτά, αλλά υπάρχει και η πολιτική πτυχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά που λέτε. Είπατε ότι υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν, ούτε να συζητήσουν για όλα τα θέματα αυτά. Αλλά όταν λέτε ότι δεν σας ακούσανε, αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την ε, αξιοπιστία της βιομηχανίας, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υγεία, τη δημόσια υγεία. Δεν είχαν υποχρέωση να τις ακούσουν αυτοί. Um, ναι, είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη μια διαδικασία να που θα μας οδηγήσει να ανακαλύψουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι μνήμες θα είναι κάπως βραχίες με την προϋπόθεση ότι το σύστημα RDE θα λειτουργήσει καλά. Θα χρειαστεί βέβαια μια περίοδος 10-15 χρόνια για να βγάλουμε τα βρώμικα δίζελ από τον δρόμο. Τι θα γίνει όμως άμα το RDE δεν είναι <clears throat> αποτελεσματικό. Αλλιώς, γιατί αν δεν είναι αποτελεσματικό όλη αυτή η διαδικασία θα μας πάει 30 χρόνια πίσω. Γι' αυτό είναι απαραίτητο αυτή τη φορά να λειτουργήσει καλά το αντί. Αν πάει καλά και υπάρχει σωστή επικοινωνία προς τους καταναλωτές, τότε θα ξεχάσουν όλοι για τα θέματα αυτά. Οι καταναλωτέ δεν του νοιάζει βέβαια όλο αυτό. Θέλουν απλώ ένα αυτοκίνητο να λειτουργεί. Θέλουν απλώ να ξέρουν ότι μπορούν να βασίζονται στι πληροφορίε που έχουν και να κάνουν τι σωστέ <clears throat> πληροφο... σωστές επιλογές για να αγοράσουν. Γι' αυτό εμείς φέρνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να μπορούν οι καταναλωτές να ξέρουν τι γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι νομίζουν ότι όλα τα diesel ευρώμικα και όλα τα Volkswagen είναι ε, τα χειρότερα αυτοκίνητα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν οι καταναλωτέ να αγοράζουν τα λάθος αυτοκίνητα επειδή είναι παραπληροφορημένοι. Χρειάζεται να υπάρξει λοιπόν μια πολιτική διαδικασία <clears throat> για να βρούμε τι έχει γίνει, ακόμα και μια δικαστική διαδικασία. Αλλά το RDE είναι η τελευταία ευκαιρία να πετύχουμε να έχουμε αυτήν την ε, διαφάνεια και νομίζω ότι το θέμα του ε, της τύπου το έχουμε προχωρήσει όσο μπορούμε. Αλλά αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά από εδώ και πέρα είναι να υπάρξει η σωστή εποπτεία των αυτοκινήτων εν χρήση. Είμαι ο επόμενος εδώ, οπότε θα κάνω την ερώτηση. Θα μιλήσω Ολλανδικά βέβαια. Κύριε Μόλντεν, Είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις για το μέλλον και να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να σας πω ότι άκουσα ότι αυτό που είπατε, ότι η φύση ακριβώς του νέου κύκλου θα βοηθήσει για να ακαλυφθούν τα κενά. Απαιτείται λοιπόν ένα υπόδειγμα δοκιμών τα οποία το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να είναι και εξελίξιμο σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. Κοιτάξτε για τα νόξ, για τα οξύδια του αζότου. Πράγματι τίθεται το θέμα του ποσοστού συμβατότητας συμμόρφωσης. Υπάρχουν ε, και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει βέβαια να προβλέψουμε για το μέλλον για να μην έχουμε αργότερα προβλήματα σε σχέση με την εκπομπή αμμονίας σαν παράδειγμα. Αν υπήρχε υπερβολική έγχυση ε, και έβγαινε αυτό από την εξάτμιση ε, ακατέργαστο, στην ουσία σημαίνει ότι καθιστούμε το ένα οξύδιο του αζότου από ένα άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσει κανείς αυτά σε πραγματική λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά και να δούμε τι δεν έχουμε προβλέψει, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις μετά και συνεχείς αλλαγές. Δεν θέλουμε οι τεχνολογίες οι οποίες απλά να σέβονται το γράμμα του RD και μετά να δημιουργούν άλλο προβλήματα. Δεν θέλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Νομίζω επίσης ότι έχουμε θέματα που δεν καλύπτει το RDE, το WLCC. Εμείς έχουμε 30% απόκληση αυτή τη στιγμή. Αυτό θα πρέπει να μειωθεί σε 15%. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, παρόλα αυτά θα υπάρχει πάντα μία διαφορά 15%. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές σε σχέση με το τι πρέπει να γνωρίσουν. Νομίζω ότι το WLTC θα έλθει στην επικαιρότητα σε λίγα χρόνια σαν θέμα συζήτηση. Είχατε επαφές σε επίπεδο οργάνωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας η Επιτροπή. Εμείς έχουμε λειτουργήσει συμβολευτικά και για το RDE και για το WLCC. Ε, ε, συμμετέχουμε δηλαδή στις διαβουλεύσεις μαζί με άλλες οργανώσεις και σώματα. Υπάρχει διάλογος δηλαδή προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε επίσης και με την GRC διάλογους. Ε, γνωρίζουν τα τεστ που κάνουμε, γνωρίζουν τα δεδομένα που συλλέγουμε και γενικά είμαστε πολύ ανοιχτοί ε, στο να συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε και είμαστε ανοιχτοί να συμμετέχουμε, να επικοινωνούμε, να βοηθάμε στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων και να καλύψουμε αυτό που ονόμασα αποτυχία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκυζίκη. Ευχαριστώ και πάλι. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι συζητήσατε τα αποτελέσματα των δοκιμασίων σας με τη Βρετανική κυβέρνηση και την, ε, της αυτο, και την αυτοκινητοβιομηχανία. Το ρώτησε και ο κύριος Έρτου, αλλά είπατε ότι δεν έχετε καθόλου ε, απαντήσεις από αυτούς. Όταν εσείς είπατε ότι υπάρχουν υπάρχει υπέρβαση τέσσερις φορές των όριων, πώς αντέδρασε η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αρχικά αποτελέσματα που δημοσίευσαν δείχναν ακόμα πιο ψηλούς παράγοντες συμμόρφωσης, 7 και παραπάνω φορές από το όριο. Όταν αρχίσαμε να τα λέμε αυτά σε συνδιασκέψεις και τα δώσαμε στις αρμόδιες αρχές η απάντηση ήταν είπαν ότι ναι, αλλά ναι, καλό είναι που μας το λέτε, αλλά δεν αντιδράσανε ουσιαστικά, δεν κάναν τίποτα. Δεν κάναν καμιά προσπάθεια να συνεννοηθούν μαζί μας. Αλλά οι εμπειρογνώμονες τους πράγματι ενδιαφερόντουσαν να μάθουν τι γίνεται αλλά δεν σημαίνει ότι στη συνέχεια μου είπανε τι θα κάνουν ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ή πώς αυτό επηρεάζει τις ε, διαπραγματεύσεις της ε, ε, Βρετανικής κυβέρνησης στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν για τα οχήματα. Αλλά πάντα θελήσανε να ξέρουμε τι λένε τα δεδομένα μας. ενδιαφέρθηκαν για τις ε, πληροφορίες αλλά δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να δώσουν περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες και να τις διαβιβάσουν στις Βρυξέλλες ώστε να αναλάβει δράση η Κομισιόν. Παραμείνανε στο νησί τους δηλαδή σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες. Είναι έτσι. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο σε όλες τις ε, συνδιασκέψεις και στην υπηρετική Ευρώπη, στη Γερμανία κυρίως, υπήρξαν ακροατήρια και πολλοί από αυτούς εκπροσωπούσαν τους Γερμανούς κατασκευαστές, τους ρυθμιστές και άλλα σώματα. Υπήρχαν και εκπρόσωποι άλλων χωρών, αλλά μικρή παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι συζητήσεις μου με τη Βρετανική κυβέρνηση ε, είναι σε εκκρεμότητα και γίνονται όταν γίνονται στα κεντρικά μας γραφεία. Κυρίως όμως έχουμε επαφές στην Γερμανία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Sono state fatte molte domande che Λοιπόν, είναι πάρα πολλέ οι ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω, αλλά έχετε δώσει πολύ καλές απαντήσεις μέχρι τώρα και γι' αυτό θα σταθώ σε κάποια υπόλοιπα. Πρώτον, εξαιρώντας τις καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων οι εκπομπές υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να θα έλεγα παρακάμπτουν την σωστή καταγραφή και να οδηγούν στην καταγραφή αποτελεσμάτων καλύτερη από την πραγματικότητα, καλύτερα από την πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το θέμα της σωστής παρακολούθησης των μετρήσεων. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Υπάρχει δυνατότητα έτσι ώστε η καταμέτρηση σε εργαστήριο και η καταμέτρηση σε πραγματική συνθήκη, έτσι ώστε διαφορετικά αυτοκίνητα να συμπεριφέρονται καλύτερα στο εργαστήριο και, καλύτερα, και χειρότερα στο δρόμο και αντίθετα άλλα καλύτερα στο δρόμο και χειρότερα στο εργαστήριο. ή μήπως παραμένει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό αν θέλετε η διαφοροποίηση ανάμεσα στο εργαστήριο και στο δρόμο. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε τώρα, δεν ξέρω αν καταλάβατε αυτό που θα ήθελα να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν σαν παράδειγμα υπάρχει μια τέτοια διαφορά σταθερή ανάμεσα στο δρόμο και στο εργαστήριο, θα αρκούσε να πολλαπλασιάσουμε με ένα συντελεστή σαν παράδειγμα τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για να δούμε ποια θα ήταν τα πραγματικά αποτελέσματα ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε ελέγχους σε εργαστήρια γιατί δεν τα κάνουμε, αλλά μπορούμε εμείς να συγκρίνουμε τα πραγματικά στοιχεία που συλλέγουμε με τα επίσημα στοιχεία που είναι εργαστηριακά. Θα απαντήσω και σε σχέση με νόξο και σε σχέση με κατανάλωση, γιατί και τα δύο είναι σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι σύντομα μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει σαφής α, ε, α, ε, ε, λόγος απόκλησης. Υπάρχουν τρομακτικές διαφορές ανάμεσα στις επιδόσεις. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που αποδίδουν εξίσου καλά ή πολύ κοντά αν θέλετε ανάμεσα στο εργαστήριο και στον δρόμο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια αυτοκίνητα χωρίς μεγάλες αποκλήσεις. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν τρομακτικές αποκλήσεις. Αν πάρουμε εμείς τα αυτοκίνητα με α κεφαλαίο στο ΕΚΟΑ, τότε προφανώς οι διαφορές είναι μικρές. Νομίζω ότι έχουμε αυτοκίνητα και στην κατηγορία α, αλλά έχουμε και στην κατηγορία H αυτά τα οποία έχουν τρομακτικές διαφορές στα 800 αυτοκίνητα που ελέξαμε στην Ευρώπη, αν θυμάμαι ότι μόνο το 1% εκπληρεί και θα έλεγα καλύπτει τα επίσημα εργαστηριακά όρια. Την 2014 ήταν μια υπανίσχυρη στον Μάρτιν. Από τότε τίποτα υπάρχουν αυτοκίνητα με τρομακτικά κενά, όπου ε, θα έλεγα η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα είναι 300% υψηλότερη από ό,τι στο εργαστήριο. Ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά, τα οποία α, έχουν τροφοδότη εξωτερικό. Υπάρχουν λοιπόν τρομερές διαφορές μεταξύ τους. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ε, ανακατασκευαστεί κάποιοι λόγοι δεδομένοι, κάποια ratio δεδομένα. Αλλά ακόμα και στο εσωτερικό αυτών των ομάδων οι διαφορές είναι τεράστιες. Λοιπόν, δεν υπάρχει ε, ενιαίος λόγος μετατροπής είτε για τα επιβατηγά είτε για τα ε, εμπορικά. Υπάρχουν τρομερές διαφορές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γοσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η παρέμβασή σας σήμερα το απόγευμα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμά σας έθεσαν το ερώτημα το οποίο θα θέσω και εγώ με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν κατανοούμε πως οι δημόσιες αρχές δεν αντέδρασαν σε αυτά τα οποία δημοσιεύσατε. Ο πρόεδρος λίγο προηγουμένως αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις κυβερνήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε σαφείς σε σχέση με αυτό. Είπατε προηγουμένως ότι προσπάθησαν να σας απαξιώσουν. Ποιος το έκανε αυτό, ποιος προσπάθησε να σας απαξιώσει και πώς. Δεν με ενδιαφέρει ε, ποιος φυσικό πρόσωπο, αλλά ήταν δημόσιες αρχές, ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σε αυτή τη φάση έγινε κάτι τέτοιο και αν έγινε πότε έγινε και πώς έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να κοιτάξει κανείς κάποιες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης. Όταν δημοσιεύουμε δεδομένα, αποτελέσματα, και όταν σαν παράδειγμα ένας κατασκευαστής για τον οποίο έχουμε δημοσιεύσει κάτι δεν είναι καλό, η αντίδραση πολλές φορές έχει σαν στόχο να μας υπονομεύσει εμάς και τη μεθοδολογία μας. Να πούνε σαν παράδειγμα ότι ο εξοπλισμός PEMS δεν είναι αξιόπιστος, ενώ εμείς γνωρίζουμε το ποσοστό ακρίβειας και αξιοπιστίας. Λοιπόν, οι κατασκευαστές και άλλοι προσπάθησαν να πούνε δημόσια μετά από ε, δημοσιεύματα ε, ότι τα συστήματά μας δεν είναι καλά και δεν ασχολήθηκαν με τα πραγματικά δεδομένα και με τα δικά μας επιχειρήματα. Και αυτά συμβαίνουν και σήμερα, λιγότερο βέβαια, αλλά συμβαίνουν και σήμερα. Προσπαθώ λοιπόν να αποφύγω κάποιες ε, ανεκδοτολογικές αναφορές αλλά θα μπορούσα από τον τύπο να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα. Ε, επίσης οι οργανώσεις οι επαγγελματικές των κατασκευαστών ε, αντιδρούν ε, αρνητικά σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουμε, ότι είναι ανακριβή, ότι κάνουμε βόλτες τυχαία και συγκρίνουμε πράγματα μη συγκρίσιμα και ότι το, τα τεστ εργαστηρίου είναι τα καλύτερα γιατί ελέγχει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία του NETC δεν βοηθούν κανέναν, είναι άχρηστα. Και μετά το Dieselgate βέβαια έχει υπέρξει μια σημαντική αλλαγή και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν αυτά τα οποία κάνουμε και συνεχίζουμε εμείς να δημοσιεύουμε στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα για δημόσιο έλεγχο. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα, αλλά σύντομα αυτό ήθελα να πω. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες και τις διαφορετικές επιχειρήσεις που κάνουν αυτά τα τεστ και ο ανταγωνισμός αυτός γίνεται με σωστό τρόπο ή στρεβλώνεται γιατί υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί σαν το δικό σας χωρίς να είναι ιδιαίτερα ανεξάρτητοι. Στην ερώτηση 12 για το ποιος χρηματοδοτεί απαντήσατε ξεκάθαρα λέγατε ότι δεν έχετε καμία εξάρτηση από έναν χρηματοδότη. Πιστεύετε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, τρευλός ανταγωνισμός με άλλους οργανισμούς που δεν έχουν αντίστοιχη με την δική σας ανεξαρτησία. I would say Θα έλεγα ότι ναι υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού, αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σύγκρουση ή τέλος πάντων μια ανάρμοστη συμπεριφορά θα το περιέγραφα ως εξή ότι η νέα, ο νέος κύκλος, το NEDC, έδωσε όμορφα στοιχεία για την αυτοκινητοβιομηχανία, κολακευτικά όσον αφορά την κατανάλωση, Τα εργαστήρια λοιπόν τα προσφέρουν αυτά, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ικανοποιημένη, οι αρχές επίσης γιατί μειώνονται τα επίπεδα ρήπανσης του εξουδίου του άνθρακος και οξυδίων του αζότου, οπότε όλοι οι παίκτες είναι ικανοποιημένοι. Οπότε τι γίνεται, οι αυτοκινητοβιομηχανίες πάνε στα ίδια εργαστήρια γιατί αυτά τους προσφέρουν, τους προσφέρουν ωραία νούμερα. Αλλά όλοι το θέλανε αυτό. Κανείς δεν ήθελε να υπάρχει ενόχληση. Αλλά δεν θα έλεγα ότι υπήρχε κακή πρόθεση. Ο κύριος Γκίζικα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Μόντεν. Είμαστε μια επιτροπή έρευνας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα πράγματα πήγαν απόλυτα σωστά ή όχι στο παρελθόν και πρέπει, θα, κάνουμε μια, θα δώσουμε μια ενδιάμεση έκθεση που θα παρουσιάσει ο κύριος Σάλμπα αλλά παράλληλα με την εργασία της Επιτροπής μας υπάρχει και η διαδικασία της ΤΑΕΚ για την εποπτεία της ε, αγοράς. Κατά τη δική σας άποψη, τι προτάσεις θα διατυπώνετε εσείς για την πράξη που, για την πρακτική πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον ώστε να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι παράνομες ε, πρακτικές, τα DVD devices κτλ. Έχετε λοιπόν κάποιες προτάσεις και για τη δική μας Επιτροπή και για την Επιτροπή της ε, Εσωτερικής Αγοράς. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Η τροποποίηση στην ε, διαδικασία έγκρισης τύπου νομίζω είναι μια σημαντική βελτίωση μπορώ να έχω μικρές ε, ε, αλλά δεν θα ήθελα εδώ να κάνω κάποια σχόλια. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να υπάρξουν αλλαγές είναι ο έλεγχος συμβατότητος εν λειτουργία του οχήματος και να μην ξεκινήσουμε μονάχα με καλές προθέσεις και σιγά σιγά να πούμε ότι ναι τα μελη πρέπει να το κάνουν και δεν θα έχουμε χρηματοδότηση εγγυημένη για αυτή τη διαδικασία και σιγά σιγά καθώς κατεβαίνει στις χώρες και σε τοπικό επίπεδο διαλύεται το σύστημα αυτό. Αυτή είναι λοιπόν η κύρια μου σύσταση πώς να επιτύχει το αντί στο μέλλον. Η δεύτερη σύστασή μου να δούμε προσεκτικά το, την κατανάλωση καυσίμων και την εκπομπή CO2 του άνθρακος γιατί δεν νομίζω το WLT θα τα λύσει αυτά και σας λέω και πάλι είναι βασικό να είναι ολιστική η διαδικασία ε, ρύθμιση των θεμάτων αυτών. Δεν είναι καλό το να έχουμε αλλού τον έλεγχο για το διοξείδιο του άνθρακος και την κατανάλωση καυσίμου και αλλού τα οξύδια ζώτου και υπάρχει και το θέμα της, ε, των, της αμμονίας που μπορεί και αυτό να αποτελέσει πρόβλημα ως ρήπος. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική λοιπόν αντιμετώπιση που δεν θα εξασφαλίσει ότι αντί να έχουμε ένα πρόβλημα θα έχουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα και αλλάζουμε ένα πρόβλημα για ένα άλλο. Να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τον έλεγχο των εκπομπών και το σύστημα να είναι έτσι ώστε η αγορά να λειτουργεί σωστά. Γιατί είναι πολύ καλά τα αυτοκίνητα τα οποία παράγονται από τη βιομηχανία και μπορούν να παραγάγουν ακόμα καλύτερα αν υπάρχει πραγματικά ισότης ανταγωνισμού και μια σαφής ρυθμιστική δομή. Νομίζω ότι μπορούν να αντιδράσουν θετικά σε αυτό το πλαίσιο. Αν έχετε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο χωρίς παραθυράκι, η προσπάθεια, γεμάτο παραθυράκι, η προσπάθεια θα πάει στο να εκμεταλλευτούν τα παραθυράκια. Η κυρία Ευχαριστώ. Θα υποφεληθώ από αυτό το δεύτερο γύρο ερωτήσεων για να παρατείνω λίγο, να συνεχίσω μετά από τις προηγούμενες ερωτήσεις μου, γιατί μου έκανε εντύπωση. Αναφερθήκατε στη στρατηγική ε, μη πιστοποίησης η καταστρατήγηση και είπατε ότι υπάρχουν και πιο περίπλοκα συστήματα πέρα από αυτά τα λογισμικά παράκαμψης ε, των προδιαγραφών. Μπορείτε να επεκταθείτε περισσότερο. Η Μιτσουμπίση στην Ιαπωνία είναι ένα καλό παράδειγμα. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ από αυτά που έχω διαβάσει και εγώ, ε, φουσκώνουν τα λάστιχα και έχουν κέρδος έτσι. Γιατί έτσι έχετε καλύτερα νούμερα όσον αφορά το σασί και γενικά έχετε χαμηλότερες εκπομπές και χαμηλότερη κατανάλωση επίσης. Για 25 χρόνια το έκαναν αυτό πριν τους τσακώσουν. Ο βαθμός από αυτό το απλό πράγμα είναι μεγάλος. Και υπάρχουν και άλλα ε, συστήματα και το TNE και άλλοι τα έχουν γράψει δεν είναι δικός μας τομέας πραγματογνωμοσύνης αυτός. Καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει από καιρούς καιρών. Πάντως λιγότερα μπορεί να κάνει κανείς το εργαστήριο για το πώς θα οδηγήσει, αν θα το κάνει αυτό με έναν έτσι πιο έξυπνο τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι στο εργαστήριο υπάρχει τέτοιο υλικό, είναι πιο περίπλοκο. Αυτά είναι απλά πραγματάκια και εκεί όπου δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν. Δεν έχει να κάνει τόσο με την παραβίαση των κανόνων, έχει κυρίως να κάνει με το ότι κάποια πράγματα δεν είναι ρυθμισμένα. Οπότε εποφελείς από αυτό το κενό και κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι όμως παράνομα αυτά καθε αυτά. Για παράδειγμα, ρωτά κυρία Ρεβό, τι δεν καλύπτεται αλλά χρησιμοποιείται ως μέθοδος. Το εύρος είναι μεγάλο. Η πίεση στα λάστιχα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και με διαφορετικά, με άζωτο για παράδειγμα, μπορείς να φουσκώσεις τα λάστιχα και να έχεις έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Ε, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με ολόκληρε μελέτες για βέλτιστες στρατηγικές. Δεν είναι δικό διά μας ε, πραγματογνωμοσύνη αυτό. Άλλοι τα έχουν μελετήσει πολύ λεπτομερέστερα και εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Πάντως αυτό το cost down test κατά τη διάρκεια επιβράδυνσης επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Όταν σκέφτονται τις δοκιμές οι άνθρωποι των οχημάτων για τα καυσαέρια, τα σκέφτονται στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια μιας πορείας. Αλλά υπάρχει και αυτή η δοκιμή στην επιβράδυνση, που δεν της δίνει το κοινό εξίσου προσοχή. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αδυναμία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Έκχαρτ, Εσείς τώρα για να κλείσουμε ο τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω, κύριε Μόλτον, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες σας τις απαντήσεις. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις που θα μπορούσα να φανταστώ. Οπότε, για να κλείσουμε. Τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το συμπέρασμά μου τουλάχιστον είναι, είναι ότι έχει να κάνει με τη ρύθμιση και δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Διορθώστε με αν κάνω σφάλμα, αλλά τα κενά εντοπίστηκαν στις ρυθμίσεις. Δεύτερον, τώρα πολλοί πολιτικοί λένε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα με τις δοκιμές RDE, δηλαδή σε πραγματική συνθήκη οδήγησης. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχτεί. Το πιο σημαντικό είναι το τέταρτο πακέτο για την ε, τελική συμμόρφωση. Οπότε ρωτάω, μια που εσείς συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουμε με το τέταρτο πακέτο. Ποιους μεγάλους κινδύνους βλέπετε από αυτό το τέταρτο πακέτο. Τι δηλαδή δεν θα κάνει για να έχουμε καθαρό αέρα και πιο καθαρά αυτοκίνητα που δεν ρηπαίνουν για να είμαστε προετοιμασμένοι τι να περιμένουμε. Η μεγαλύτερη κίνδυνη είναι Η κάθε χώρα είναι αυτή που θα δει πώς θα προχωρήσει, οπότε μπορεί μερικές φορές να μην γίνουν καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το EPA και το Board της Καλιφόρνια κάνει εποπτικούς ελέγχους, αλλά ούτε και αυτοί δεν βρήκαν το πρόβλημα με τη Volkswagen. Μια μη κυβερνητική οργάνωση το βρήκε. Και το EPA στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, παρόλο που διαθέτει εξοπλισμό, κόσμο κτλ, υποχρηματοδοτείται. Αλλά δεν χρειάζονται πολλοί πόροι για να ελέγξει κανείς αρκετά αυτοκίνητα ώστε να μπορεί να διαπιστώσει ποιος κλέβει. Οπότε το θέμα είναι ότι συμφωνηθεί να τεθεί σε εφαρμογή και να συνοδεύεται από την κατάλληλη χρηματοδότηση. Δεύτερον, ναι, όντως, η ρύθμιση είναι το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ότι για όλα αυτά η, ρύθμιση, η έλλειψη ρύθμισης, θα έλεγα ότι εδώ υπήρχε μια ευχάριστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παικτών στον τομέα αυτό και χρειάστηκε μια εξωτερική δυναμική παρέμβαση για να ε, χαθεί αυτή η ισορροπία. Δεν ήταν θέμα τεμπελιάς, δεν ήταν θέμα προθυμίας. Για πολλούς λόγους το υπάρχον σύστημα εξακολουθήσε να υπάρχει, γιατί από αυτό εποφελόνταν πολλοί. Και όλοι θέλανε να διατηρήσουν το, τους ελέγχους αυτούς στα εργαστήρια, οπότε έκαναν τα πάντα για να παραμείνουν αυτοί οι έλεγχοι στα εργαστήρια. Οπότε έχει να κάνει με τις χώρες μέλη, με την αυτοκινητοβιομηχανία. Όλοι οι παίκτες έχουν κάποιο βαθμό ευθύνης για την κατάσταση. Όλοι βολεύονταν αφήνοντας τα πράγματα ως είχαν, για να μην ξυπνήσει το τέρας. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε ο κατάλογο ομιλητών, οπότε θα ολοκληρωθεί έτσι και η ακρόασή μα, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο προσκεκλημένου μα, και τον κύριο Κάου και τον κύριο Μόλντεν, για τη συμμετοχή σα εδώ. Τώρα, οι συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλουν επιπλέον ερωτήσει γραπτά μπορούν στη γραμματεία μέχρι την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη 23 του μηνός. Το μόνο που έχω να σας πω ακόμα είναι ότι αύριο το πρωί συνεχίζουμε 21 Ιουνίου στις 9 το πρωί με ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την έκθεσή μας την προσωρινή και με εκπροσώπους από τις αρχές τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ.